Θα ήθελα να σας καλωσορίσω σε αυτή την εργομήγυρη προκειμένου να βοηθήσουμε την Κομισιόν να ασχοληθεί με την αναδιατύπωση της Οδηγίας 2201 του 2003 σχετικά με την διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση των αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέρημνας, ο οποίος κατοργείται με τον οργανισμό 1347-2000. Υπάρχουν πολλοί διακεκριμένοι συνάδελφοι εδώ, συμπεριλαμβανομένου και του Σαντέου Σουσιάφκα εισηγητή και ο αρμόδιος από την Κομισιόν, η αρμόδια συγγνώμη, και Κάρεν Φαντριχαχόβεν. Α, ναι, ναι, εδώ στο βάθος είναι. Είσαστε πρόσδεκτοι λοιπόν όλοι σας στην Επιτροπή μας. Έχουμε καλέσει επίσης μέλη από την Επιτροπή Αναφορών, την Επιτροπή Γυναικών που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το ζήτημα. Καλώς ορίζω και τον, την Αντιπρόεδρο κυρία Μαγκίνες, αρμόδια για θέματα διαφορών γονικής μέρημνας, προσθέσεων παιδιών κλπ. Με οποία δίνει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ που με καλωσορίσατε, μου δώσατε δυνατότητα να μιλήσω εδώ. Ευχαριστώ όλους όσους συμμετείχαν στις εργασίες για αυτό το σημαντικότατο θέμα. Εν είδη εισαγωγή σχετικά με το τι κάνουμε, είναι στην ιδιωτική σφαίρα που γίνεται αυτή η δουλειά, προσωπικού χαρακτήρα, ασχολούμεθα με άτομα, με ανθρώπους, με γονείς που δεν μπορούν να καταλήξουν σε κάποιες διευθετήσει και συμφωνίες και ζητούν βοήθεια. Καμιά φορά μπορούμε να βοηθήσουμε, άλλες όχι. Υποθέτω ότι αυτά είναι θέματα που θα πρέπει να συζητήσουμε σε αυτή τη δουλειά που κάνουμε. Είναι προσωπικό αυτό το θέμα και καμιά φορά ε, υπάρχει σύγκρουση μεταξύ νόμου και προσωπικών πτυχών. Και καμιά φορά δεν συμφωνούν διάφορα μέρη, οπότε πρέπει να δούμε ποιο είναι το συμφέρον το καλύτερο των παιδιών. Πολλές φορές στην παρουσίασή μου εγώ αναφέρω το συμφέρον των παιδιών και δεν ζητώ συγγνώμη γι' αυτό, θα το αναφέρω επανειλημμένα στην εργομή γυρί μας. Είναι πολύ σημαντικό να πω στους ενήλικες ότι τα παιδιά είναι δική μας ευθύνη, δεν είναι ιδιοκτησία μας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για το πώς ε, βλέπουμε τις ρυθμίσεις ε, και πώς ε, προστατεύουμε το συμφέρον τους. Από πολλές πλευρές τα κράτη-μέλη προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το θέμα με αποτελεσματικό τρόπο. Σε πολλές περιπτώσεις όμως δεν καταλήγουν σωστά οι προσπάθειες για τους ενδιαφερομένους και αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη. Το πρώτο θέμα που αφορά το πρόβλημα της απαγωγής των παιδιών. Είναι τόσο σοβαρό το γεγονός. Στο γραφείο μου ξέρουμε ότι υπάρχουν κάποια παιδιά τα οποία δεν μπορούμε να βρούμε, δεν ξέρουμε που βρίσκονται. Καμιά φορά η απαγωγή των παιδιών είναι προσωρινό φαινόμενο και λύνεται εύκολα το πρόβλημα. Αν πράνε κακά τα στραβά τα πράγματα, οι συνέπειες είναι καταστροφικές για τα παιδιά, για τον γονέα που έχει μείνει πίσω, για τις οικογένειες, για τους παππούδες και έχει αντίκτυπο για μια ολόκληρη ζωή και πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε τρόπους να ελαχιστοποιήσουμε αυτό, αυτά τα σοβαρά αποτελέσματα. Ε, καμιά φορά είναι δύσκολο να διελευκάνουμε τις καταστάσεις και έχουμε δικαστές, επαγγελματίες που έχουν κάθε καλή πρόθεση και αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες λεπτομέρειες συναισθηματικού χαρακτήρα αλλά αληθεύει επίσης ότι μπορούμε να σκληρύνουμε εργαζόμενοι από ε, τις πολλές υποθέσεις που εξετάζουμε, σκλίνουμε κάπου και πρέπει να το δούμε αυτό. Λοιπόν, είναι ένα γενικό εργαλείο ε, ε, για την οικογένεια και οι δικαστές και οι νομικοί δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τα πολύ δύσκολα οικογενειακά ζητήματα. Ούτε τα δικαστήρια ίσως είναι ο καλύτερος χώρος για την αντιμετώπιση αυτών των πολύ ευαίσθητων ζητημάτων και ίσως και να είναι και πιο δαπανηρή λύση, να το λάβουμε και αυτό υπόψη το κόστος. Είναι σημαντικό να έχουμε υπόψη ότι οι μακροσκελείς δικαστικές διαδικασίες όσον αφορά τη γονική ευθύνη μπορούν να αυξήσουν ε, τις εντάσεις και αυτό δεν βοηθά κανέναν. Ε, πολύ συχνά είναι καλύτερα να προσπαθήσουμε να έχουμε μια ατμόσφαιρα επίλυσης αξιοπρεπούς του προβλήματος σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα και να μην κρατάει πολλή ιστορία. Καμιά φορά όμως ε, τελικά χάνουμε τον έλεγχο του χρόνου Πρέπει να παραδεχτούμε ότι τα νομικά συστήματα των κρατών εδράζονται επί παραδοσιακής νοοτροπία και ότι υπάρχουν διαφορές και οι διαφορές πρέπει να εξεταστούν. Λοιπόν, έχουμε διάφορες συγκεκριμένε περιπτώσεις με υπέρ και κατά, αλλά όλες είναι υποθέσεις που αφορούν ανθρώπινη τραγωδία, κυρίω για τα παιδιά. Και ξεπερνάνε οι συνέπειε στην άμεση οικογένεια. Και γι' αυτό είμαι πεπισμένη ότι πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στη διαμεσολάβηση και την ενδεχόμενη εμπλοκή κοινωνικών υπηρεσιών και ψυχολόγων. Σύστημα υποστήριξης πρέπει να υπάρχει και να είναι πολύ ισχυρό. Ακόμα και όταν δύο άνθρωποι πολεμούν, έχουν αποξενωθεί και δεν μπορούν να καταλήξουν σε συμβιβασμό και φτάνουν στο σημείο να βλέπουν τι καταστροφικέ συνέπειε για το γονέα που μένει πίσω και για το παιδί και πάλι θα ήταν δυνατόν και τότε και πρέπει να το εξασφαλίσουμε, να του επιβληθούμε, να μπορέσουμε να τους κάνουμε να συνομιλήσουν μέσω διαμεσολαβητή τα δύο μέρη. Η διαμεσολάβηση δεν εφαρμόζεται μόνο σε αυτό το τομέα τη νομοθεσία, αλλά και σε πολλού άλλου. Πρέπει να βοηθήσουμε τον κόσμο λοιπόν να καταλάβει ότι η διαμεσολάβηση μπορεί να αποτελεί πραγματικά μια καλή λύση και ίσως αυτό θα πρέπει να το κουβεντιάσουμε ανοιχτά στην κοινωνία ούτως ώστε αν προκύψει για οποιονδήποτε από εμά ένα πρόβλημα στη ζωή μας να μην θεωρούμε σαν πρώτη επιλογή τα δικαστήρια αλλά τη διαμεσολάβηση και ίσως το νομικό σύστημα σαν ε, μια διέξοδο για επίλυση του προβλήματος. Η διαμεσολάβηση για μένα είναι σημαντική και θετική εναλλακτική ε, έναντι της ε, νομικής ε, διαμάχης και ελαχιστοποιείται η ένταση και για τα παιδιά και για τους γονείς, τους ίδιους. Η διαμεσολάβηση δίνει χώρο και χρόνο για αποτελεσματική επικοινωνία και νομίζω ότι η αποτελεσματική επικοινωνία είναι κάτι που όλοι χρειαζόμαστε εκπαίδευση σε αυτό. Όσον αφορά την επίλυση των συγκρούσεων σε οικογενειακές περιστάσεις, δεν υπάρχει επαρκή επικοινωνία και η διαμεσολάβηση μπορεί να δώσει αυτό το χώρο και το χρόνο για επικοινωνία. Επίσης μπορεί να βοηθήσει στην αποφυγή προβλημάτων, να προλάβουμε προβλήματα. Αυτή πρέπει να είναι η προσέγγισή μας, ώστε να μην δημιουργηθούν αυτές οι καταστάσεις όπου ακολουθείται η χείριστη επιλογή, απάγεται ε, το παιδί από το σπίτι του και το πηγαίνουν σε άλλο κράτος μέλο, ή και σε χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Πρέπει αυτό να το έχουμε όλους ιδιαίτερους υπόψη. Τώρα, για τις φιλικές διευθετήσεις. Αυτό θα θέλαμε όλοι για να ελαχιστοποιούμε τα προβλήματα για όλους. Τούτου λεχθέντος, η νομοθεσία όμως θα πρέπει να εφαρμόζεται, οπότε θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τους νόμους, τους κανονισμούς, ούτως ώστε να έχουμε αποτελεσματικό νομοθέτημα που βασίζεται επί των εμπειριών μας. Παραδέχομαι ότι υπάρχουν αυτές οι περιπτώσεις που η δημοσιολάβηση δεν μπορεί να ισχύσει, να εφαρμοστεί. Πρέπει να δοκιμαστεί, αλλά αν δεν μπορεί να λειτουργήσει και να συμφωνήσουν τα εμπλεκόμενα μέρη, τότε βεβαίως πρέπει να είμαστε λογικοί και ευαίσθητοι και να δούμε πώς μπορεί να παρέμβει ο νόμος. Πρέπει να επεξεργαστούμε το θέμα της επικοινωνίας και της δικτυώσεως των δικαστικών συστημάτων να επικοινωνούν μεταξύ τους οι δικαστές. Αυτό συμβαίνει σε πολλές περιπτώσεις, αλλά μπορεί να βελτιωθεί. Η εκπαίδευση, η κατάρτιση, θα επαναλάβω αυτή τη λέξη κατάρτιση, διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να συντονιστεί ο κόσμος με αυτή την πτυχή και το ανθρώπινο δυναμικό και την ομοθεσία. Πρέπει να σκεφτούμε όλα αυτά τα θέματα και να εντοπίσουμε τρόπους με τους οποίους μπορούμε να βοηθήσουμε τους πολίτες διαφυλάσσοντας τα συμφέροντα των παιδιών. Ότι καμιά φορά όταν η σύγκρουση είναι πολύ έντονη, δεν βλέπουν οι εμπλεκόμενοι τα παιδιά, δεν ακούνε τα παιδιά και ίσως το παιδί δεν λαμβάνεται καν υπόψη. Και πρέπει να δώσουμε στα παιδιά ε, ένα ασφαλές περιβάλλον στο βαθμό του δυνατού, ούτως ώστε να διατηρείται και μια σχέση και με τους δύο γονείς, αν είναι δυνατόν αυτόν. Όχι μόνο με εκείνον που έχει μείνει πίσω, αλλά και με τους δύο γονείς κυρίως όταν ζουν οι γονείς κάτι κράτη-μέλη. Θα πρέπει να ε, δημιουργούνται διάφορες συμφωνίες και να εφαρμόζονται συμφωνίες. Ίσως αυτό θα πρέπει να εξετάσουμε, την εφαρμογή, την υλοποίηση, τον, την εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων. Ο κανονισμός Βρυξέλλες 2α υπήρξε επιτυχής. Αυτό βοήθησε τους πολίτες Ευρωπαϊκής Ενώσεως, δημιουργώντας ευρύ φάσμα αναγνωρίσεων αποφάσεων, επιβολή αποφάσεων στον ευαίσθητο τομέα που αφορά τα παιδιά, τι γονικέ ευθύνε. Επίση, διευκόλυνε τη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και των κεντρικών αρχών των κρατών μελών και συμπλήρωσε την σύμβαση για την απαγωγή παιδιών, για την επιστροφή των παιδιών και να αποτραπεί μελλοντική απαγωγή παιδιών. Για το θέμα τώρα των κεντρικών αρχών υπάρχει και ένα βασικό ρόλο για τι κεντρικέ αρχέ να παρέχουν οι αρχές αυτές έγκαιρα πληροφορίες στο ίδιο το κάτω μέλος, αλλά να συνεργάζεται η αρχή αυτή και με άλλα κράτη-μέλη και πρέπει να ενισχυθούν οι δεσμοί μεταξύ των αρχών, των φορέων και των μελών, τα δύναμη δεσμοί αυτοί. Πολύ συχνά βλέπετε ο γονέα, κυρίω αν δεν μένει στο κάτω μέλο που είναι η πατρίδα του και του πάρουν το παιδί του ενό γονιού, ε, θα αντιμετωπίσει αυτό ο γονιό που έχει μείνει πίσω κρίση. Και χρειάζεται πληροφορίε. Εύκολη πρόσβαση στι πληροφορίε. Δεν πρέπει να παλεύει για να βγάλει άκρη και να βρει βοήθεια. Καλωσορίζω λοιπόν την αλλαγή που υποβάλλεται στην πρόταση για να τη οδηγία του κανονισμού που διευκολύνει τι διαδικασίε επιστροφή των παιδιών. Δημιουργείται το, η βάση για να ακούγεται η άποψη του παιδιού. Βασικό αυτό, το κάνουν αυτό κάποια κάτι μέλη με καλό τρόπο και πρέπει να δούμε πώ η φωνή του παιδιού μπορεί να ακούγεται και με αποτελεσματικό τρόπο. Χρειάζεται η βελτίωση των διασυνοριακών εκτελέσεων των εντολών επιστροφή και θα πρέπει να εξασφαλίσει τη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και μεταξύ των κεντρικών αρχών αυτών. Και το υπογραμμίζω αυτό. Η επανάληψη καμιά φορά λειτουργεί, διότι ο κόσμο τελικά θα το λάβει το μήνυμα. Επίση, καλωσορίζω τη ρητή εισαγωγή στο άρθρο 23, παράγραφο 2, συμπληρωματικού βήματο τη διαδικασία, όπου τα δικαστήρια απαιτείται να καλούν τα μέρη, ούτω ώστε να συμμετάσχουν στη μεσολάβηση του ταχύτερο δυνατόν, διότι είναι προ το βέλτιστον όφελο του παιδιού να εξευρεθεί μια συμπεφωνημένη λύση. Γι' αυτό ο των κεντρικών αρχών για την παροχή των πληροφοριών που ανέφερα είναι κρισίμου σημασία. Συνοπτικά λοιπόν, πριν το γεύμα συναντήθηκα με εκπροσώπους του γραφείου μου ε, και που αναλαμβάνουν τα μέλη του γραφείου μου διάφορες υποθέσεις και είναι πολύ ευαίσθητα ε, τα μέλη αυτά σε διάφορες υποθέσεις. Πολλές υποθέσεις υποβάλλονται σε εμά πολύ αργά και όπως σας είπα η έγκαιρη επέμβαση είναι πάρα πολύ σημαντική. Άρα πρέπει αυτά τα θέματα να αντιμετωπιστούν με ευαίσθητο τρόπο με μεγάλη ευαισθησία για τους εμπλεκομένους. Είναι πρόκληση και για τις διεθνείς οικογένειες. Πρέπει να φροντίσουμε να βοηθούμε τον κόσμο σε εποχές που το χρειάζονται, όπου οι σχέσεις καταραίουν. Επιλογές υπείας νομοθεσίας μαζί με την πιο σκληρή νομοθεσία πρέπει να ταιριάζουν και να συμπληρώνονται και πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη επανειλημμένα τη φωνή του παιδιού και τα δικαιώματα του παιδιού. Προσβλέπω λοιπόν στις εργασίες των οποίων θα ηγηθεί ο εισηγητής μας που θα εξετάσει λεπτομερώς ε, τον κανονισμό και την αναδιατύπωση του κειμένου και το τμήμα πολιτικής ε, το ευχαριστώ που διοργάνωσε αυτή την ε, συνεδρία σε αυτό το εργαστήριο και ευχαριστώ και το υπηρεσία έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εξέτασε την εξολόγηση συνεπιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στρέφομαι προς τον Ρόμπερτ και τους συναδέλφους του της γραμματείας ε, μας ε, που πάντα μας βοηθούσαν όταν χρειαζόμαστε τη βοήθειά τους, την υποστήριξή τους και τον προσανατολισμό τους αντιμετωπίζοντας ευαίσθητα νομικά θέματα τα οποία είναι ζητήματα που αφορούν την καρδιά μας και θέματα θλιμμένων καρδιών. Άρα είναι πολύ ευαίσθητα ζητήματα αυτά, αλλά και πολύ δύσκολα και σκληρά πλευρά νομική. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Μαρή, που ήρθες και αυτά τα αρχικά σου σχόλια. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν το πρώτο σημείο, την παρουσίαση της προτάσεως περί αναδιατυπώσεως. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Κάρεν Βαντεκέρ Κρεχόβε της Γενικής Διευθύνσεως Δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να μας παρουσιάσει τις βασικές πτυχές της προτάσεως περί αναδιατυπώσεως και έχετε ένα εικοσάλεπτο στη διάθεσή σας. Thank you, Chair. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και Καλησπέρα σε όλους. Είναι μια χαρά να βρισκόμαστε εδώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που διοργανώσατε αυτό το εργαστήριο. Και θα ήθελα να ευχαριστήσουμε και τον κύριο Σβιεύκα, ο οποίος ήταν εισηγητής για το θέμα αυτό και το οποίο έδωσε το έναυσμα για την κίνηση της εργασίας ε, στο Κοινοβούλιο μέσω αυτού του εργαστηρίου. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω την πρόταση της Επιτροπής και πολλές από τις ε, πτυχές της πρότασης ήδη έχουν ε, διευκρινιστεί, έχουν παρουσιαστεί από την κυρία Μακίνες. The regulation just... Ο κανονισμός, για να δούμε περί τίνος πρόκειται, ασχολείται μόνο με διασυνοριακά θέματα, σημαντικά διασυνοριακά θέματα, όπως είπε η κυρία Μακίνες, και αφορά την ε, αναγνώριση της δικαιοδοσίας ε, μεταξύ χωρών μελών και την εφαρμογή αποφάσεων σε τρία ζητήματα. Ε, θέματα που αφορούν διαζύγια και χωρισμούς, θέματα γονεϊκής ευθύνης θέματα κυδαιμονίας και θέματα πρόσβασης στο παιδί και ζητήματα απαγωγής παιδιών. Αυτό είναι το πλήρες ε, εύρος του κανονισμού. Ο κανονισμός αυτός έχει εφαρμοστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση πάνω από 20 χρόνια και ξεκινήσαμε μια διαδικασία αξιολόγησης ε, τουλάχιστον πριν από δύο χρόνια. Και το έργο το οποίο κάναμε στην ε, ε, βάση της ε, προπαρασκευής της αναθεώρησης του κανονισμού ε, ήταν, διαμορφώθηκε ως εξή. Είχαμε μια δημόσια διαμούλευση το 2014, της οποίας προηγήθηκε η σύνταξη μιας, η έκθεση μιας, έκθεση εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και βεβαίως ε, αυτό έφερε πολλά στοιχεία, πολλές πληροφορίες. Στη συνέχεια ε, ασχοληθήκαμε με την υπάρχουσα νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και τα πολλά ερωτήματα και αναφορέ που έγιναν από πολίτες στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και κάναμε επίση μια μελέτη αξιολόγηση, είχαμε μια ομάδα εμπειρογνωμόνων ε, των διαφόρων ε, διαφερόμενων ούτε ώστε να συντηθεί η λειτουργία και είχαμε, ε, η οδηγία συγγνώμη, και είχαμε και ε, τις συναντήσεις ε, με διαφόρους παράγοντες και όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία συλλέξαμε μας επέτρεψε να καταλήξουμε σε ορισμένα συμπεράσματα. Το βασικό συμπέρασμα ήταν ότι ο κανονισμός πραγματικά λειτουργήσε καλά, άρα μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία επιδέχονται περαιτέρω βελτιώσεων και προσπαθήσαμε να επικεντρώσουμε την προσοχή μας σε αυτά τα θέματα. Τα θέματα αυτά ήταν τα πιο επίγοντα ε, και αφορούσαν κυρίως την ε, ευθύνη των, ε, των γονέων στις διεθνείς περιπτώσεις απαγωγών. Προσπαθήσαμε λοιπόν να επικεντρώσουμε την προσοχή μας στα θέματα αυτό βάζοντας ε, Βάζοντα στην άκρη θέματα διαζυγίων κλπ. Και εδώ ε, αναζητήσαμε τα έξι βασικά, τους έξι βασικούς τομείς της ε, περιπτώσης, διεθνής περιπτώσης απαγωγών, το, το να ακούμε το παιδί, την, την κατάργηση, την κήρυξη της εκτελεστότητας, την ε, ε, τοποθέτηση των παιδιών διασυνοριακά σε άλλες ε, χώρες μέλη. Αυτά είναι τα βασικά σημεία και υπάρχουν και κάποια άλλα τα οποία δεν είναι λιγότερο σημαντικά αλλά παρόλα αυτά είναι κάπως λάσονα αν θέλετε και για παράδειγμα, ήδη η κυρία Μακίνες ε, ανέφερε την πρόθεση της διαμεσολάβησης στο παρόν ε, πλαίσιο του κανονισμού. Και για να έρθουμε εν συντομία στις προταθήσεις βελτιώσεις, ε, θα ήθελα να πω τα εξή. Η πρώτη σχετίζεται με τις διεθνείς παγωγές παιδιών. Ο βασικός στόχος των βελτιώσεων είναι να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα ε, της ε, διαδικασίας, νομικής διαδικασίας και η επιτάχυνση. Ε, γιατί εάν είναι χρονοβόρες αυτές τις διαδικασίες, τότε η επιστροφή του παιδιού πολύ συχνά δεν έχει πλέον κανένα αντικείμενο. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά να μην γίνονται όμοιρα, να μην εγκλωβίζονται σε χρονοβόρες νομικές διαδικασίες οι οποίες οδηγούν σε μη αναστρέψιμες επιπτώσεις αυτό ε, οδήγησε στην ε, πρόταση του να γίνουν κάποιες βελτιώσεις ούτως ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες. Ε, καταρχήν θα έπρεπε να διευκρινιστούν οι προθεσμίες τις εντός των οποίων θα έπρεπε να ληφθούν οι αποφάσεις επιστροφής των παιδιών. Και προσπαθήσαμε να μειώσουμε το μέγιστο, τη μέγιστη διάρκεια εντός της οποίας θα πρέπει να γίνει η επιστροφή του παιδιού. Αυτή τη στιγμή η περίοδος αυτή είναι 165 μέρες το διάστημα κατά το οποίο συνήθως επιστρέφεται το παιδί. Ε, εμείς προτείναμε 18 εβδομάδες, δηλαδή 1,5 μήνα, ε, που ότι είναι μια αποδεκτή προθεσμία. Προσπαθήσαμε επίσης να μειώσουμε τον αριθμό των δικαστηρίων ε, στα οποία παρουσιάζονται τα παιδιά γιατί δυστυχώς οι τέτοιες διεθνείς περιπτώσεις απαγωγών παιδιών ε, δεν είναι κάτι που πάει στα δικαστήρια καθημερινά και η τεχνική πολυπλοκότητα μεταξύ των διαφόρων νομικών οργάνων δεν είναι απλό θέμα. Άρα λοιπόν ε, θα πρέπει οι διαδικασίες να είναι πολύ πιο απλές ε, στην περίπτωση που υπάρχουν αρμόδια δικαιοδοτικά όργανα για αυτές τις ε, πολύ συγκεκριμένε και ε, εξαιρέσεις ελπίζουμε περιπτώσεων και γι' αυτό θέλουμε να περιορίσουμε τον αριθμό των δικαστηρίων σε κάθε χώρα που θεωρούνται αρμόδια για να εκδικάσουν αυτές τις υποθέσεις απαγωγής παιδιών σε πολλές χώρες μέλη υπάρχει η δυνατότητα να γίνουν αλλεπάλληλες ε, εφέσεις οι οποίες ε, καθυστερούν ακριβώς την επιστροφή του παιδιού. Γι' αυτό θέλουμε να περιορίσουμε το πιθανό αριθμό των εφέσεων από τη μία και να διασφαλίσουμε ότι τα δικαστήρια στις χώρες μέλη μπορούν να εξασφαλίσουν την ε, εκταλιστότητα των αποφάσεων ούτω ώστε να μπορεί άμεσα να επιστραφεί το παιδί. Αυτές είναι οι βασικές αλλαγές ε, τις οποίες ε, προτείναμε ε, όσον αφορά αυτές τις περιπτώσεις απαγών των παιδιών σε διεθνή κλίμακα. Το δεύτερο θέμα αφορά την ακρόαση του παιδιού, το οποίο επισημάνθηκε επίσης από την κυρία Μακίνες και προς το συμφέρον του παιδιού βεβαίως είναι ένα βασικό στοιχείο ε, στοιχείο κλειδί για τον κανονισμό, το συμφέρον του παιδιού και η δυνατότητα κρόασης του παιδιού. Και βλέπουμε από την ε, λειτουργία του κανονισμού ότι οι διάφοροι τρόποι μέσα των οποίων ε, ακούγονται τα ίδια τα παιδιά στις διάφορες χώρες μέλη δημιουργούν δυσκολίες σε διασυνοριακό επίπεδο και αυτό δημιουργεί κάποια εμπόδια στην αναγνώριση και στην εφαρμογή δικαστικών αποφάσεων στο εξωτερικό. Προσπαθούμε λοιπόν να εισαγάγουμε στον ίδιο τον κανονισμό μια υποχρέωση για τα δικαστήρια να ακούσουν το παιδί. Η υποχρέωση αυτή ήδη είναι κατοχυρωμένη στην Διεθνή Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, αλλά θα θέλαμε να συμπεριληφθεί και να εφαρμόζεται σε όλες τις νομικές διαδικασίες ε, που αφορούν τον κανονισμό για το παιδί. Άρα να ενισχυθεί αυτή η πτυχή του να ακούγεται το παιδί και το δεύτερο στοιχείο είναι οι διασυνορικές επιπτώσεις αυτής της ακρόασης. Δηλαδή θέλουμε να εξασφαλίσουμε χώρες μέλη αμοιβαία να αναγνωρίζουν τα εθνικά συστήματα της κάθε χώρας για την ακρόαση των παιδιών. Άρα, εάν η ακρόαση διεξάγεται με έναν τρόπο διαφορετικό από ό,τι θα γινόταν στη δική σας χώρα, για παράδειγμα, παρόλα αυτά, αυτός δεν θα πρέπει να είναι λόγος για μια απόρριψη μια αναγνώριση της απόφασης ε, στη δική σας χώρα, αλλά θα πρέπει να υπάρχει μια ελεύθερη διακίνηση των δικαστικών αποφάσεων. Το δεύτερο, το επόμενο σημείο αφορά ακριβώς ε, την, αυτή καθ' αυτή η ελεύθερη ε, διακίνηση ε, των δικαστικών αποφάσεων, άρα δηλαδή την κήρυξη εκτελεστότητας και υπάρχουν και άλλοι κανονισμοί στους οποίους ήδη έχει γίνει αυτή η κήρυξη εκτελεστότητας εξ ολοκλήρου ή εν μέρη για ορισμένε αποφάσει για παράδειγμα στα δικαιώματα πρόσβαση και σε ορισμένε αποφάσει που αφορούν την επιστροφή του παιδιού. Έχει ήδη εφαρμοστεί αυτό, αλλά θα θέλαμε να διευρύνουμε αυτή την αυτόματη αναγνώριση και εφαρμογή, δηλαδή την άμεση κήρυξη τη εκτελεστότητας σε όλε τι αποφάσει που αφορούν ε, την επιστροφή των παιδιών, ε, δηλαδή ε, αποφάσεις για επιστροφή των παιδιών. θε, θέλουμε βεβαίως να εισαγάγουμε εδώ τις αναγκαίες ασφαλιστικές δικλίδες, ούτως ώστε να παράσχουμε μια επαρκή προστασία, ε, για παράδειγμα, της ε, υποχρέωσης νομικής παράστασης. Το δεύτερο σημείο, το οποίο ήδη αναφέρθηκε από την κυρία Μακίνης, αφορά την ε, παρούσα ε, εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων. Γιατί αυτό είναι το, η βασική δυναμία η οποία, ε, στην οποία επιδρώσαμε την προσοχή μας στην δημόσια διαβούλευση και αφορά την ισχύουσα, την εφαρμογή όσο έχει μέχρι στιγμής. Το ενωσιακό δίκαιο μέχρι στιγμή έχει επιδρώσει την προσοχή του στην αναγνώριση μιας της απόφασης και την ε, εφαρμογή στην άλλη χώρα. Αλλά το πώς ακριβώς εφαρμόζεται αυτή η δικαστική απόφαση, αυτό επαφιέται στην ευχέρεια των χωρών μελών και δεν προβλέπεται μια συγκεκριμένη ε, διαδικασία για ε, θέματα ακριβώ οικογενειακά. Είναι ίδια όπω και σε νομισματικά οικονομικά θέματα. Άρα λοιπόν, εδώ ε, δεν λαμβάνεται υπόψη τι ανάγκες να υπάρξει μια πολύ ταχεία διαδικασία στην περίπτωση των παιδιών. Και αυτό συνιστά πραγματικό, ένα πραγματικό εμπόδιο όσον αφορά τη διακίνηση, την αναγνώριση δηλαδή, να μπαίνει αναγνώριση των δικαστικών αποφάσεων και την ε, επιστροφή των παιδιών. Γι' αυτό θεωρούμε, στο πλαίσιο της αναδιατύπωσης, είναι σημαντικό να ε, να δούμε πώς μπορεί να παλευθεί αυτό το εμπόδιο της ε, πρόσβασης κατά βάση στην ε, δικαιοσύνη. Προτείνουμε λοιπόν να υπάρξει μία νομική ασφάλεια σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την αναγνώριση των δικαστικών αποφάσεων για τις απαγωγές των παιδιών. Και επίσης θέλουμε να περιορίσουμε την ε, προθεσμία της εφαρμογής των δικαστικών αποφάσεων. Θεωρούμε ότι θα έπρεπε να, να ισχύει το διάστημα των ε, έξι εβδομάδων για την εφαρμογή της δικαστικής απόφασης και αν η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να τηρηθεί, τότε θεωρούμε ότι το δικαστήριο θα έπρεπε να είναι σε θέση να εξηγήσει γιατί δεν μπόρεσε να γίνει η εφαρμογή της απόφασης εντός της προθεσμίας των έξι εβδομάδων. Το επόμενο σημείο στο οποίο προτείνουμε αλλαγέ αφορά την τοποθέτηση του παιδιού σε μια άλλη χώρα μέλος και αυτό αφορά καταστάσεις όπου για παράδειγμα το παιδί θα πρέπει να τοποθετηθεί ε, σε μία ανάδοχο οικογένεια, σε μία άλλη χώρα ή σε κάποιο ίδρυμα. Ε, πρόκειται λοιπόν για αυτό το είδος ε, διασυνοριακής τοποθέτησης του παιδιού. Ε, και υπάρχει το άρθρο 56 το οποίο ασχολείται με το θέμα αυτό και λάβαμε πολλές ε, προτάσεις από ανθρώπους που εργάζονται ακριβώς στο θέμα αυτό της διασυνοριακής τοποθέτησης του παιδιού επισημένοντας ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα όσον αφορά την αποτελεσματικότητα αυτή τη τοποθέτηση του παιδιού διασυνοριακά. Υπάρχουν πολλέ καθυστερήσει. δεν υπάρχει επαρκή νομική ασφάλεια στο θέμα αυτό και τα παιδιά εγκλωφίζονται σε γραφειοκρατικές διαδικασίε, ενώ πολύ συχνά ε, τέτοιου είδου καταστάσει είναι πραγματικά κατεπίγουσες γιατί το παιδί θα πρέπει να το φροντίσουν συχνά σε μια άλλη χώρα μέλη, μέλος. Γι' αυτό προσπαθήσαμε να πετύχουμε μια ενιαία διαδικασία σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτως ώστε να υπάρχει αυτή η ενιαία διαδικασία για τις τοποθετήσεις των παιδιών και πάλι μια προθεσμία και πάλι 8 εβδομάδων ε, για το μέλο, ε, μέλος προς το οποίο υποβάλλεται η αίτηση να την αποδεχθεί ή να την απορρίψει. Και τέλος, η συνεργασία μεταξύ των κεντρικών αρχών, θέμα το οποίο ήδη έχει επισημανθεί και που είναι πραγματικά οι βασικές ε, αρχές ε, στον κανονισμό αυτό, γιατί υποστηρίζουν το έργο του δικαστού όσον αφορά τη λειτουργία του κανονισμού και πολύ συχνά είναι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι ε, σε άμεση επαφή με τους γονείς. Προκειμένου να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των κεντρικών αρχών, προτείναμε να διευκρινιστεί και να ενισχυθεί ο ρόλος του στο κείμενο του κανονισμού, ούτως ώστε να γίνει σαφέστερο τι ακριβώς αναμένουμε από αυτούς όταν ε, ε, υποβάλλονται αυτές οι αιτήσει και προτείναμε, το είπε η Μακίνες, να συμπεριφερθούν στο σύστημα συνεργασίας και η, το σύστημα, και η κοινωνική λειτουργή. Πολύ συχνά είναι αναγκαίο να υπάρχουν κάποιες ε, αναφορές, κάποιες εκθέσεις σε σχέση με την ακριβή κατάσταση του παιδιού, που μπορεί να αναλάβουν το παιδί που θα, το, που θα τοποθετηθεί και κατά πόσο ε, πληρώνονται όλες ε, οι συνθήκες για την ε, παρκή φροντίδα του παιδιού. Άρα θα πρέπει οι κοινωνικοί λειτουργοί να συνεργάζονται με τις κεντρικές αρχές. Αυτά είναι τα έξι βασικά, οι έξι βασικοί τομείς της αναθεώρησης. Υπάρχουν κάποιες άλλες ε, λάσονες ε, αλλαγές ε, στις οποίες δεν θα αναφερθώ εγώ αλλά νομίζω ότι τις εντοπίσετε εσείς στις συζητήσεις σας. So, thank you Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση. Προτού να προχωρήσουμε, θα ήθελα να καλωσορίσω την κυρία Γκέπχαρντ, πρώην διαμεσολαβητή για θέματα απαγωγών τέκνων. Περνάμε λοιπόν στο επόμενο ζήτημα. Καλωσορίζω τον κύριο Μίλος Χάπτκα, Χάτκαπα, κάπως έτσι. Πρόεδρο της ομαδας βιξελες Βιξέλλες 2α και για την αναδιατύπωση αυτής. Έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου, κυρίε και κύριοι. Η Σλοβακική Προεδρία παρακολούθησε τις εργασίες ε, σχετικά με την αναδιατύπωση αυτού του κανονισμού διότι θέλουμε να ε, θέσουμε τις προτεραιότητες μας ε, θέλουμε τις προτεραιότητες μας αυτό ζήτημα. Η Σλοβακική Προεδρία ανέκαθεν την ιδιαίτερη σημασία σε αυτόν τον κανονισμό αφενός διότι ήταν το πρώτο μέσο στον χώρο της δικαστικής συνεργασίας που εφαρμόστηκε στην Σλοβακία συγχρόνως με τα υπόλοιπα μέλη της Ένωσης. Όλα τα άλλα ε, εργαλεία ε, τέθηκαν σε εφαρμογή μετά την ένταξη της Σλοβακίας. Ο δεύτερος λόγος ε, υπήρξε ότι ε, καταλάβαμε ότι υπήρχε ανάγκη να γίνει αυτό, διότι ε, χρειαζόμαστε συνεργασία των υπολοιπών μελών, διότι ήμασταν, ε, συμμετείχαμε στην συνθήκη του 86, σύμβαση του 86, και πολλές διατάξεις σε αυτή την ε, οργανισμό έχουν εφαρμοστεί. Μόλις διαπιστώσαμε λοιπόν ότι η Κομισιόν πρόκειται συντόμως ε, να αναλάβει πρωτοβουλίες μετά από την έναρξη της προεδρίας μας να διατυπώσαμε τις ε, προτεραιότητες μας ε, προκειμένου να έχουμε έχουμε δυνατότητα να συμβάλλουμε και εμείς στο έργο αυτό, ειδικά στο ζήτημα του περιβάλλοντος. Γιατί το περιβάλλον, διότι θεωρούμε ότι αυτός ο φάκελος, αυτό το ζήτημα, είναι πολύ περίπλοκος και ευαίσθητος δεν είναι διόλου απλό διότι θα πρέπει να εγκριθεί ομόφωνα από το Συμβούλιο και ένα καλό περιβάλλον εργασιακό που θα επιτρέψει στις αντιπροσωπείες να συζητήσουν σε βάθος και ανοιχτά ε, τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους θα οδηγούσε σε ένα αποτέλεσμα το οποίο μπορεί να επιτευχθεί σε μεταγενέστερο χρόνο και το οποίο θα αντανακλά τις επιθυμίες και τις προσδοκίες όλων των κρατών μελών. Κατά τη διάρκεια της Σλοβαϊκής Προεδρίας ε, είχαμε πέντε συναντήσεις ε, σε τεχνικό επίπεδο. Η ε, πρώτη διεξήχθη πριν από τις θερινές διακοπές και επικεντρώθηκε επί των έξι ζητημάτων τα οποία η Κάραν αναφέρε και περιλαμβάνει την πρόταση της Κομισιόν, όπως επίσης και την ε, αξιολόγηση επιπτώσεων. Οι επόμενες ε, συναντήσεις ε, εξέτασαν τις επιμέρους διατάξεις του κειμένου με χρονολογική σειρά και έχουμε προς το παρόν εξετάσει τα τρία πρώτα κεφάλαια και η τελευταία συνάντηση που διεξήχθη το δεκαημέρο μας οδήγησε στο να αρχίσουμε το δέτημα της, αναγνω... της αναγνώρισης και της επιβολής. Γενικά, η θέση των εψοποιών είναι υπέρ κάτω μάλλον ήταν της προτάσεως του, καλωσορίζουμε την δυνατότητα και την ευκαιρία που προσφέρεται για την επίλυση πρακτικής φύσης αλλά και νομικής φύσης προγράμμα, ε, ε, ζητημάτων που αντιμετωπίζουν οι αρχές αλλά και οι πολίτες κατά τη διάρκεια αυτής της δεκαετούς περίοδου εφαρμογής του κανονισμού. Καταλαβαίνετε ότι πρόκειται για την πρώτη εξέταση του εγγράφου και οι συζητήσεις αφορούν ιδιαίτερα στην διευκρίνηση των διατάξεων και την κατανόηση του κειμένου αυτών των διατάξεων. Πολλοί εκπρόσωποι στους οποίε εκφράζονται με, την, με κάποιες επιφυλάξεις διότι δεν έχουν ακόμα οριστικοποίηση τις, ε, τις ε, διαδικασίες και τις συζητήσεις στο εσωτερικό τους. Οι προτάσεις της Κομισιόν και των κρατών μελών οδηγούν σε μια εκτενή ανταλλαγή απόψεων αναφορικά με το πώς κάποιες λύσεις μπορούν ή δεν μπορούν να λειτουργήσουν σε ορισμένα νομικά συστήματα. Δεδομένου του πρώιμου ακόμα σταδίου, είναι αδύνατον να προβλέψουμε ενωσδήποτε ενδείξεις για το πώς θα ε, ε έχει στο μέλλον ο νοοκανονισμός οποιοδήποτε λοιπόν αναφορά μου ενδεχομένα να στείλει ένα, ένα σφαλμένο μήνυμα. Αυτό το οποίο όμως μπορώ να σας πω χωρίς να σας ε, να σας παρασύρω σε παρανοήσει, είναι κάποια πράγματα τα οποία μπορούν να σε εκπλήξουν, άλλα μπορεί να όχι. Τέλο, εκτός από κάποια πράγματα λοιπόν τεχνικής φύσης αναφορικά με το πω είναι, ε, διατύπωση θα επηρεάσει τις υφιστάμενε πρακτικές ε, ορισμένες ορισμένε πω πως οι ε, νέε διατάξεις θα επηρεάσουν τις διαδικαστικές ε, αυτονομίες των κρατών μελών και ποιες θα είναι οι επιπτώσεις αυτών των διατάξεων και στις εσωτερικές διαδικασίες σε ό,τι αφορά τώρα τα πιο συγκεκριμένα ζητήματα θα αναφερθώ σε κάποια από αυτά μία συζήτηση ήταν η αντικατάσταση του όρου court, δικαστήριο, με τον όρο authority, αρχές. Ακόμα και τώρα στο τρέχον το υφιστάμενο έγγραφο το όρος ε, δικαστήριο αφορά τις αρχές. Υπάρχουν κάποιες διαφωνίες ε, μεταξύ των οποίων ότι αυτές οι αλλαγές θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σοβαρές ε, παρανοήσεις και γι' αυτό πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί σχετικά με το ποιες διατάξεις θα πρέπει να εφαρμόζονται μόνο στα δικαστήρια κόρτς και όχι σε άλλες αρχές οθόρητης. Τώρα σχετικά με το πεπετσουάτσιο φόρη, σου ευθυγράμμιση ε, του κανονισμού στον, ε, στον ε, της Χάγης έχει διάφορα υπέρ και κατά. Η ιδέα του να επεκταθεί η δυνατότητα για τους διάδικους για τους διαδίκους ε, διευρύνοντας το χρονικό διάστημα το οποίο αυτή η επιλογή μπορεί να επιτευχθεί δημιουργεί κάποια ζητήματα τα οποία αφορούν την πρακτική εφαρμογή αλλά και τις συνέπειες μιας τέτοιας παρα... χρονικής παράτασης. Το νέο άρθρο που ε, προβλέπει μέτρα προστασίας και που περιλαμβάνεται στην ε, σύμβαση της Χάγης του 1986 οδήγησε σε μακροσκελείς ε, συζητήσεις αλλά δημιούργησε και μια σειρά από ερωτήματα και ζητήματα όπως αυτά τα οποία αφορούν στο ζήτημα της απαγωγής ε, του τέκνου και την αναγνώριση και επιβολή παρομοίων μέτρων. Το, το ζήτημα των άλλων, το, άλλων ε, θεμάτων ε, να, χρειάζεται μάλλον να συζητηθούν περαιτέρω για το πώς αυτή η πολιτική θα πρέπει να αντανακλάται στο κείμενο του κανονισμού. Η διάταξη για το δικαίωμα του τέκνου να εκφράζει την άποψή του ή την άποψή τη θεωρήθηκε ότι θα πρέπει να ε, συμπεριληφθεί, ότι καμία αντιπροσωπεία δεν ε, αμφισβητεί την ε, σημασία αυτής της αρχής. Τώρα, σχετικά με το νέο κεφάλαιο για την απαγωγή τέκνων, οι αντιπροσωπείες καλωσόρισαν την νέα δομή, διότι κρίνουν ότι το θέμα της απαγωγής θα πρέπει να έχει ένα δικό του κεφάλαιο, να αφιερωμένο σε ένα κεφάλαιο. Τώρα, σε σχέση με τις ισχύουσες διατάξεις, αλλά επίσης ε, προέκυψαν και μια σειρά από πρακτικής φύσης ερωτήματα, ορισμένε από τις οποίες ε, ανέφεραν την ανάγκη για περισσότερη φιλοδοξία η οποία θα πρέπει να εμπνεύσει αυτές τις νέες διατάξεις. Κατά τη διάρκεια της Λουβαϊκής Προεδρίας, δύο ακόμα συνεδριάσεις της ομάδας θα ε, διεξαχθούν για την εξέταση του κεφαλαίου 4, αναγνώριση και επιβολή και η σημαντική ζήτηση ε, βρίσκεται ακόμα ενώπιον μας. Κρίνοντας ε, από, από αυτά τα οποία μας έχουν δηλώσει οι μπορώ να καταλήξω πιστε, ε, ότι έχουμε πετύχει το, το, το, στο σχέδιό μας. Το κλίμα είναι πολύ καλό, ανοιχτό και επικοδομητικό στην ομάδα εργασία. Είμαι βέβαιος ότι οι επερχόμενες προεδρίες θα συνεχίσουν τις συζητήσει στο αυτό πνεύμα και θα μας οδηγήσει σε μια επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων. Ευχαριστώ για την προσοχή σα. Mr. Ευχαριστώ κύριε Χατάπκα. Ευχαριστώ για αυτά που μας είπατε και για την όλη επισκόπηση της καταστάσεως για τα τεκτενόμενα στην ομάδα εργασίας σας. Μπορούμε να ξεκινήσουμε λοιπόν τις συνεδριάσεις μας. Τη σύνοδος, η πρώτη σύνοδος ασχοληθεί διαθρωμένη διαδικασία επιστροφής παιδιών σε σχέση με την απαγωγή παιδιών. Δεύτερο τμήμα, αύξηση συνεργασίας μεταξύ κεντρικών και δικαστικών αρχών. Τμήμα τρίτον, οι κρίκοι που μας λείπουν. Ξεκινάμε με το πρώτο τμήμα λοιπόν. Καλωσορίζω θερμά την δόκτωρα Ηλιάρα Μπρτέλη από το Ελβετικό ε, Ινστιτούτο Συγκριτικού Δικαίου Δώστε μας την άποψή σας για την διατύπωση του κανονισμού Βρυξέλλες 2α για παγωγή και επιστροφή παιδιών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για το προνόμιο, την τιμή και τη μεγάλη χαρά να παρίσταμε. Αυτή η χαρά συνοδεύεται και από συνέστημα ευθύνης, διότι είμαι απόλυτα πεπισμένη ότι το νομοθέτημα που συζητούμε σήμερα μπορεί να επηρεάσει κατά πολύ το μέλλον της ενώσεως και τον τομέα ελευθερίας, δικαιοσύνης και ασφαλείας. Διστάζω κάπως λέγοντας αυτές τις λέξεις, γιατί περνάμε φρικτές εποχές, τρομακτικές εποχές. Όλοι βλέπουμε πως ο Ευρωπαϊκός Χώρος Ελευθερίας, Δικαιοσύνης και Ασφαλείας δεν μπορεί να θεωρηθεί σαν κάτι δεδομένο, δεν είναι ένα δόγμα, εξαρτάται από τα συναισθήματα των Ευρωπαίων πολιτών για την πρόσβαση σε αυτή την ελευθερία δικαιοσύνη και ασφάλεια εντός των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως αφορά τη δυνατότητά τους να προστατεύσουν τα παιδιά τους εντός αυτών των συνόρων Είχα το προνόμιο να παρουσιάσω εδώ το 2014 μια μελέτη του Ελβετικού Ινστιτούτου Συγκριτικού Δικαίου που εκεί τονίζαμε την ανάγκη να προωθηθεί η κατάρτιση των δικαστικών μέσω της γνωστοποίησης των ξένων νομικών συστημάτων και των ξένων γλωσσών. Όλα αυτά τόσο ώστε να βαθυνθεί και να ενισχυθεί ένας κοινός, μια κοινή ευρωπαϊκή δικαστική κουλτούρα που είναι προϋπόθεση για δύο στόχους. Ομαλή συνεργασία σε διαδικασίες επιστροφής και συναφείς διαδικασίες και γρήγορη νομική σταθεροποίηση της καταστάσεων αφορά το παιδί που εμπλέκεται σε αυτού του είδους τις υποθέσεις. Καλωσορίζω την επιτευθύσα πρόοδο μέσω της αναδιατυπώσεως, όμως πρέπει να γίνουν και άλλες προσπάθειες ευαισθητοποίησεως. Θα παρουσιάσω αυτά τα βήματα, υπενθυμίζοντας κάποια απλά στοιχεία. Το πρώτο. Ένας κοινό ευρωπαϊκός νομικός πολιτισμός υπάρχει στην πράξη, στην καθημερινή ρουτίνα των Ευρωπαίων πολιτών. Προσελκύει ανθρώπους από άλλα μέρη του πλανήτη. Δεν είναι μόνο προνόμιο ειδικευμένων νομικών εμπειρογνωμόνων όπως εμείς. Το ζούμε καθημερινά. Δεύτερον, ένας ευρωπαϊκός νομικός πολιτισμός μπορεί να τροποδοτηθεί από το Ιους Κομούνε με την ελεύθερη διακίνηση καθηγητών, ερευνητών όσον αφορά τις κοινέ βάσεις που έχουμε πολύ συχνά θεωρώ καταχρηστικό και προσβλητικό να στιγματίζουμε νομικές πράξεις ή τη μεταφορά της κατοικίας του παιδιού ή την απαγωγή του παιδιού. Είναι σημαντικό να μην υποτιμούμε το βάρος των λέξεων. Στο σημείωμά μου σας δίνω τρία παραδείγματα γονικών συμπεριφορών που ίσως να μπορούν να χαρακτηριστούν ως απαγωγές παιδιών. Πρώτη περίπτωση. Δύο ελβετοαιγυπτιακά κορίτσια που πήγαν στην Αίγυπτο για δύο εβδομάδες με τον πατέρα τους για διακοπές και χάρη σε δικαστική άδεια του Ελβετικού Δικαστηρίου του Κουν παρά την αντίσταση της μητέρας των κοριτσιών. Η μητέρα τώρα μαζεύει μέσω φιλανθρωπίας τα χρήματα προσπαθώντας να επιστρέψουν τα παιδιά που έχει στην κυδαιμονία της στην Ελβετία. Τα παιδιά δεν πηγαίνουν σχολείο στην Αίγυπτο και οι Αιγυπτικές αρχές δεν γνωρίζουν που βρίσκονται. Όπως ξέρετε η Αίγυπτος δεν έχει κυρώσει τη σύμβαση του 1998 και η συνεργασία μεταξύ Ελβετίας και Αιγύπτου δεν έχει κατάλληλες δομές. Δεύτερη υπόθεση παιδί αυστριανού ζευγαριού που είχαν σχέσεις αποστάσεως μέχρι ότου να είναι τριών ετών το παιδί. Τελικά η μητέρα αποφάσισε να πάει στο σύντροφό της για να μεγαλώσει το παιδί στην Αυστραλία και με τους δύο γονεί. Εκατέψει τη δουλειά της και πήγε να κατοικεί στην Αυστραλία. Ανακάλυψε όμως εκεί ότι ο φίλο της είχε σχέσεις με άλλες γυναίκες και αποφάσισε να τα μαζέψει και να επιστρέψει στη Βρετανία. Ζήτησε να γυρίσει ο πατέρας στη Βρετανία, να μεταφέρει το παιδί στην ε, Βρετανία. Μονομερή ήταν η απόφαση για το που θα μείνει το παιδί από τη μητέρα και δεν συμφωνούσε ο πατέρας. Δεν ενεγκρίθη η επιστροφή, διότι το παιδί ποτέ δεν είχε διαμείνει μόνιμα στην Αυστραλία. Διότι η μητέρα κατάλαβε ότι ο εταίρος της είχε άλλες σχέσεις τρεις μέρες μετά που πάτησε το πόδι της στην Αυστραλία. Τρίτη υπόθεση διάλυση μιας λιθωνικής οικογένειας. Το παιδί 9 ετών. Έπρεπε το κορίτσι να ζήσει με τη μητέρα της, χωρίς επαφή με τον πατέρα. Όμως, η μητέρα την έφερε στην Αγγλία. Προσπάθησε να βρει δουλειά εκεί. Ο παλιάς ζήτησε να επιστραφεί το παιδί στην Αγγλία και το αγγλικό δικαστήριο διέταξε την μητέρα να επιστρέψει το παιδί στη Λιθουανία εκτός αν μπορούσε να παραστεί να πάρει άδεια από το δικαστήριο στη Λιθουανία να επιστρέψει στην Αγγλία. Τι μας λένε αυτές οι υποθέσεις. Πρώτον, for... υποθέσεις όπως η πρώτη είναι υποθέσεις για την οποία η Σύμβαση της Χάγης του 1998 είχε σχεδιαστεί. Ο, όταν τα παιδιά θεωρούνται σαν ιδιοκτησία κατά την άποψη κάποιου γονιού. Αυτή η αντίληψη απορρέει από ερμηνεία προσωπικών δικαιωμάτων που απορρέουν από νομική νοτροπία και που κάποια δικαιώματα αποδίδεται συγκεκριμένο φίλο. Δηλαδή, αλλά έχει συγκεκριμένα δικαιώματα ο πατέρα, συγκεκριμένα η μητέρα. Και υπάρχει σύγκρουση μεταξύ των νοτροπιών και των ευρωπαϊκών αρχών. Και αυτή η σύγκρουση θα πρέπει να αποτρέπει άλλα τέτοια φαινόμενα στον ευρωπαϊκό χώρο ελευθερίας, δικαιοσύνης και ασφάλειας. Λαμβάνοντα υπόψη αυτό, ο Ευρωπαίος νομοθέτης ίσως θα πρέπει να δώσει μεγαλύτερη προσοχή στα φαινόμενα που αφορούν ευρωπαϊκές υποθέσεις. Ευρωπαϊκές υποθέσεις μοιάζουν μόνο σε κάποιο βαθμό με την απαγωγή παιδιών Αυτές οι υποθέσεις σχετίζονται άμεσα συχνά με τη θεμελιώδη ελευθερία μετακίνησης εργαζομένων, όπως το είδαμε στην τρίτη υπόθεση. Σε πρόσφατη απόφαση του ΔΕΚ, 27 Οκτωβρίου, το δικαίωμα ελεύθερης μετακίνησης ανθρώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν έχει αντίκτυπο στη ζωή παιδιού, θεωρείται ότι αν επηρεάζεται η μία άμυα απόφαση για μετακίνηση, επηρεάζει αρνητικά τη ζωή του παιδιού, ε, πρέπει να εξετάζεται. Δηλαδή επηρεάζει το δικαίωμα μετακίνηση του γονιού, ότι αυτή την περίπτωση. Το άρθρο 13 της Σύμβασης της Χάγης χρησιμοποιείται για την απαγόρευση επιστροφής του παιδιού σε αυτές τις περιπτώσεις. Η απόφαση επιστροφής του παιδιού ίσως να παραβιάζει κάποια θεμελιώδη δικαιώματα κάποιου γονέως. Όπως και η απόφαση επιστροφή, όπως και μη επιστροφή μπορεί να επηρεάζει δικαιώματα γονιού. οποίο έχει ζήσει διάλυση οικογένεια. ξέρει τα προβλήματα, πώς να υπάρχει κατάλληλο περιβάλλον να μεγαλώσουν τα παιδιά μου αφού αποτύχει η οικογένεια. Ακόμα και σε απλές περιπτώσεις. Χρειάζεται να αναδιοργανωθεί η οικογένεια, να βρει δουλειά, να, κανονίσει τα οικονομικά. Λέει ο πρόεδρος λίγο πιο σιγά. Um, είναι και θέμα οικονομικό, πως θα τακτοποιηθεί το οικονομικό όταν διαλυθεί η οικογένεια. Πρέπει να εξετάζουν ποια είναι η κατάσταση που αφορά το παιδί. Αν αδιατυπωθεί ο κανονισμός και γίνει αυτό που λέει η κυρία Μαγκίνες και αν συμβάλλει στο να μειωθούν οι ανθρώπινες τραγωδίες η αναδιατύπωση αυτή τόσο το καλύτερο. Θέλουμε να ακούγεται η φωνή του παιδιού. Αυτό είναι το σημαντικό. Και αυτό με τη βοήθεια διαμεσολάβησης. Για να διαφερθούν οι διαμεσολαβητές στην υπόθεση. Τα δικαιώματα του παιδιού που προστατεύονται από τον ΑΙΕ δεν θέλουμε να αποτελούν πάρα πολύ βαριά ευθύνη για κάποιο γονιό. Πρέπει να υπάρχει αμοιβαία εμπιστοσύνη. Και αυτό να γίνει μέσω διαλόγου. Να υπάρχει διάλογο με του γονεί και το παιδί, μέσω διαμεσολαβητών. Με τη συμβολή κεντρικών αρχών. Μέσω ανταλλαγή πληροφοριών. Αυτά πρέπει να ενισχυθούν. Πρέπει να ερευνάτε κατάλληλα υπόθεση πριν ληφθεί απόφαση για την κυδαιμονία του παιδιού. Χρειάζεται ευρύ πλαίσιο όταν εξετάζουμε την κάθε υπόθεση. Και όταν κάνουμε και την αδιατύπωση του κανονισμού. Είναι η ύψη της σημασίας. Και πρέπει να βλέπουμε ε, πόσο ενταγμένος είναι ο κάθε γονιός στη χώρα που ζει το παιδί. Ας πούμε ότι μετακινείται ένας γονιός για να κάνει οικογένεια. Και ξαφνικά δεν πάει καλά η ιστορία, διαλύεται η οικογένεια και βρίσκεται ξεκρέμαστος ένας γονιός, δεν ξέρει τη γλώσσα, δεν έχει δουλειά, δεν έχει επαφές. Χρειάζεται βοήθεια τότε. Βασικός παράγων για να μην αισθανθεί ο ένας γονιός ότι έχει απομονωθεί στη χώρα στην οποία μετανάστευσε. Και αυτή πρέπει να είναι η φιλοσοφία τη ανδιατύπωσης. Χρειάζεται στενή συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκομένων φορέων όσον αφορά τι υποθέσει απαγωγή παιδιού. Κεντρικέ αρχέ, δικαστέ, επαγγελματίε, διαμεσολαβητέ, κοινωνική λειτουργή κλπ. κλπ. Και κυρίω οι γονεί. Χρειάζεται συντονισμένη λύση, συνενετική. Και θα την αποφασίζει ο δικαστή τη χώρα συνήθου διαμονή του παιδιού. σε επαφή με την χώρα νέας διαμονής του παιδιού. Εκ των υστέρων έτσι θα δημιουργείται αμοιβαία εμπιστοσύνη και θα αποδίδεται δικαιοσύνη στους Ευρωπαίους πολίτες. Αυτά είχα να σας πω, σκεφτείτε τα. So, thank you very much and, and so... Ευχαριστώ, πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Συγγνώμη που σας διέκοψα, αλλά πάντοτε γίνεται αυτό όταν δεν μπορεί να ακολουθήσει η διερμηνία τον ομιλητή. Ναι, λοιπόν, ας... Ας σκεφτούμε λοιπόν τη σημασία των όσων μας είπατε. Ε, και τώρα θα καλέσουμε τον Κρίστοφ Πάουλ, ε, διαμεσολαβητή στο Διεθνές Κέντρο Διαμεσολάβησης σε οικογενικές συγκρούσεις και περιπτώσεις απαγωγής των παιδιών. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε τη δυνατότητα να σας μιλήσω και να μοιραστώ μαζί σας κάποιες ιδέες που αφορά διασυνοριακές περιπτώσεις οικογενειακής διαμεσολάβησης τη δεκαετία του 90 του περασμένου αιώνα θέματα οικογενειακών διενέξεων που αφορούσαν την κυδαιμονία των παιδιών έδωσαν το έναυσμα στην γαλλική και γερμανική κυβέρνηση να προωθήσουν ζητήματα διαμεσολάβησης. Ε, Γάλλοι και Γερμανοί συνεργάστηκαν, ένας Γερμανός και ένας ε, Γάλλος ε, βουλευτής ε, συνεργάστηκαν ε, εκπροσωπώντας τους δύο ακριβώς αυτούς πολιτισμούς και οι δύο μιλούσαν και τις δύο γλώσσες και οι δύο μιλούσαν και γαλλικά και γερμανικά και εκπροσωπούσαν και τα δύο φύλλα γιατί ήταν άνδρας και γυναίκα αντιστοίχως. Αυτή λοιπόν, η, αυτό το γαλλογερμανικό project ε, διαμεσολάβησης αποτέλεσε το πυρήνα της μετέπειτα ε, εξέκλησης. Και το μοντέλο αυτό υιοθετήθηκε στη συνέχεια και κάτω από το πρίσμα άλλων άθρων της Σύμβασης της ε, Χάγης διαπιστώνουμε ότι οι κεντρικές αρχές θα πρέπει να λάβουν όλα τα δεδεγμένα μέτρα για να εξασφαλίσουν την εκούσια επιστροφή του παιδιού ή να οδηγήσουν σε μια φιλική διθέτηση ε, του θέματος. Ε, η Σύμβαση των 96 της Χάγης αναφέρει ρητά τη χρήση της διαμεσολάβησης της ε, συνδιαλλαγής και άλλων μέτρων, όχι μόνο για περιπτώσεις απαγωγής παιδιών, αλλά για πάσης φύσεως ε, διασυνοριακές οικογενειακές ε, υποθέσεις που αφορούν την γονεϊκή ευθύνη και την τοποθέτηση των μεταφορά των παιδιών. Ε, τώρα με τον ε, ε, κανονισμό των Βρυξελών το δικαστήριο θα πρέπει να εξετάζει κατά πόσο τα ενεχόμενα μέρη είναι πρόθυμα να αποτανθούν σε μια, να χρησιμοποιήσουν μια διαδικασία διαμεσολάβησης ε, εφόσον με, υπό την προθόθεση να μην, αυτό, να μην επιφέρει αυτό μια καθυστέρηση της διαδικασίας. Όπως είπε η κυρία Μακίνες, ε, ζητήματα παγωγών ε, παιδιών ε, σηματοδοτούνται από μια ιδιαίτερος ευαίσθητη δυναμική των σχέσεων και αποτελούν πολύ σύνθετα ζητήματα. Σε πολλές περιπτώσεις η διαμεσολάβηση είναι η, πρώτη, η μόνη ενδεδειγμένη λύση γιατί ακριβώς ε, λαμβάνει υπόψη και τις συναισθηματικές και τις νομικές πτυχές του ζητήματος, της σύγκρουση. Οι διασυνοριακοί διαμεσολαβητές μπορούν να λειτουργήσουν σαν γέφυρα μεταξύ των γονέων. Οι διαμεσολαβητές δεν θα πρέπει μόνο να έχουν γενικές εξαιρετικές επικοινωνικές δεξιότητες, αλλά και ειδικέ γνώσεις στο πεδίο της διαπολιτισμικής επικοινωνίας και επίλυση συγκρίσεων ένας διαμεσολαβητής με καθαρά νομικό υπόβαθρο δεν έχει συνήθως τέτοιου είδους επικοινωνικές δεξιότητες. Ταυτόχρονα η διαμεσολάβηση σε διασυνοριακές περιπτώσεις γίνεται πάντοτε κάτω από τη σκιά του νόμου, γιατί ο νόμος εκπροσωπεί ένα σημαντικό πλαίσιο στις περιπτώσεις αυτές, η σημασία του οποίου δεν μπορεί να ε, ενδεχομένω μπορεί να υποτιμηθεί από διαμεσολαβητέ που δεν έχουν ακριβώ αυτό το νομικό υπόβαθρο. Σε περιπτώσει ε, διεθνών απαγών των παιδιών, ε, το χρονικό πλαίσιο ασκεί τρομερή πίεση, γιατί η διαμεσολάβηση θα πρέπει να γίνει άμεσα και δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε καθυστερήσεις. Γι' αυτό ε, κάναμε ένα μοντέλο εκπαίδευσης για τους ε, διαμεσολαβητές και η εκπαίδευση αυτή έχει δημορφωθεί ως εξής. Ε, αφορά και τις δύο κουλτούρες των γονέων. Οι διαμεσολαβητές δηλαδή πρέπει να γνωρίζουν και τους δύο, τις δύο διαφορετικές κουλτούρες, να μιλούν και τις δύο γλώσσες και θα πρέπει να έχουν νομικό και ψυχοδυναμικό υπόβαθρο ε, και θα πρέπει να εκπροσωπούν και τα δύο φύλλα. Βάσει τη δική μου εμπειρία, θα μπορούσα να πω ότι για την επιτυχία πολλών ε, διασυνοριακών περιπτώσεων, στι οποίε εγώ έχω διαμεσολαβήσει, ακριβώ αυτό το μοντέλο της ε, κοινής, ε, της διπλής διαμεσολάβησης ήταν, είναι το πιο ενδεδειγμένο προκειμένου να οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα. Ε, υπάρχει ένα δίκτυο διαμεσολαβητών και όπως βλέπετε έχουμε πάνω από 450 ειδικευμένους διαμεσολαβητές οι οποίοι έχουν την έδρα του στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε ολόκληρο τον κόσμο και διαμεσολαβούν σε πολλές ε, γλώσσες. Δεν υπάρχουν αρκετά στατιστικά στοιχεία όσον αφορά τις διασυνοριακές οικογενειακές υποθέσεις οι οποίες ε, καταλήγουν στην διαμεσολάβηση. Η ΜΙΚ, ο οργανισμός ε, στον οποίο εγώ αναφέρομαι, είναι ο μόνος ο οποίος δημοσιοποιεί στατιστικά στοιχεία που αφορά διασυνοριακές περιπτώσεις οικογενειακής διαμεσολάβησης και ε, λαμβάνει τις πληροφορίες από την υπηρεσία συμβουλευτικής και διαπιστώνεται μια τεράστια αύξηση ε, τα τελευταία χρόνια ε, όπου υπήρχαν ε, τον τελευταίο χρόνο ε, πάρα πολλές αιτήσεις, πάνω από 600 αιτήσει διαμεσολάβησης. Γνωρίζουμε από αιτήματα και από το feedback που είχαμε από τους διαμεσολαβητές ότι οι αριθμοί αυτοί αντανακλούν μόνο το ίμιση του πραγματικού αριθμού των διαμεσολαβήσεων. Οι διασυνοριακές υποθέσεις υποβάλλουν αίτηση ε, στο ΜΙΚ, ε, δημοσιοποιούνται στον ιστότοπο, αλλά μπορούν επίσης να υποβάλουν μία αίτηση στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο, ε, το οποίο αναφέρθηκε εδώ. Άρα υπάρχουν γονείς οι οποίοι απευθύνονται άμεσα στους διαμεσολαβητές χωρίς να περάσουν από το συμβουλευτικό όργανο του ΜΙΚ. Ε, τα στατιστικά στοιχεία αναφέρονται στι σημειώσεις μου. Ε, είχαμε ε, 2015 έγιναν ε, ε, έρευνε. έρευνες σε 15 χώρες, έγιναν έρευνες από γονείς, από μητέρες, από πατεράδες και από κρατικές αρχές κυρίως από τις Ηνωμένε Πολιτείε, από τη Γαλλία, την Πολωνία, το Βέλγιο, το Ηνωμένο Βασίλειο, το Μεξικό, την Τουρκία κλπ. Στο τελευταίο πίνακα βλέπουμε τον αριθμό των διεθνών αιτήσεων για διαμεσολάβηση. Και εδώ σημαντικό είναι ότι η στατιστική δείχνει μια σημαντική αύξηση περιπτώσεις επανατοποθέτησης των παιδιών. Ε, μέχρι τώρα έχουμε ε, το 2016-26 περιπτώσεις και είναι ε, και βλέπουμε ότι οι γονείς γνωρίζουν όλο και περισσότερο ότι το παιδί εφόσον ε, περάσει από αυτή τη διαδικασία τελικά θα επιστραφεί. Ε, και δείχνει αυτό ότι οι υπηρεσίες ε, προκαταρτικής πριν από την διαμεσολάβηση είναι ο παράγον κλειδί για να φτάσουν, να αποτανθούν οι γονείς και να, σε εμά και να ζητήσουν, να αποβάλουν έτσι αυτή τη διαδικασία υπάρχει ένα 65% των διαμεσολαβήσεων ε, της ΜΙΚ που τελικά καταλήγουν σε μια ικανοποιητική ε, πλήρως ή εν μέρη ε, ικανοποιητική διαμεσολάβηση. Και αφορούσαν οι περιπτώσεις 242 παιδιά. Ε, θα ήθελα να ολοκληρώσω με δύο συστάσεις. Η εκπαίδευση για τους δικαστές στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να διευκολυνθεί σε σχέση με το πώς να ενθαρρυνθούν τα ενεχόμενα μέρη να ξεκινήσουν αυτή τη διαδικασία το νωρίτερο δυνατό ε, και θα πρέπει οι διαμεσολαβήσεις ε, να γίνονται χωρίς ε, περιττές καθυστερήσεις. Οι αρχές θα πρέπει να ενθαρρύνουν τα ενδιαφερόμενα μέρη να ξεκινήσουν τη διαδικασία παράσχοντας πληροφορίες έχουμε στον ιστότοπό μας κάποια τέτοια στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τα δικαστήρια. Η εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων θα πρέπει να γίνεται άμεσα και θα πρέπει να διευρυνθεί η εφαρμογή αυτών των αποφάσεων και πέραν των ορίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, ε, ε σας έδειξα έναν υπολογισμό. Υπάρχει μια μείωση κατά δύο τρίτα του κόστους και αυτό δείχνει ποιο είναι το οικονομικό όφελος των ε, διασυνοριακών διαμεσολαβήσεων. Γιατί ο παράγον κόστος εδώ είναι πολύ καθοριστικός. Άρα οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, θα πρέπει να ενθαρρύνονται να προχωρήσουν σε τέτοιου είδους διαδικασίες διαμεσολάβησης. Οι δημογραφικές μεταβολές στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως αποτέλεσμα των πρόσφατων μεταναστευτικών ροών οδήγησαν σε μία αύξηση τέτοιων διανέξεων περί κυδαιμονία των παιδιών όταν δεν υπάρχει, εφόσον δεν υπάρχει ένα διεθνές πλαίσιο. Και σε αυτές τις περιπτώσεις η διαμεσολάβηση είναι ο μόνος τρόπος να επιληθούν αυτές οι διανέξεις μεταξύ των γονέων και θα ήθελα να σας απευθύνω τη σύσταση να διευκολυθούν όλα τα προγράμματα εκπαίδευσης ούτως ώστε να υποστηριχθούν οι διαδικασίες διαμεσολάβησης και να υπάρξουν και ειδικευμένοι λειτουργοί. Ευχαριστούμε πολύ. Και για το, να κλείσουμε το πρώτο, το τελευταίο, το, το πρώτο τμήμα μάλλον η δόκτωρ Νικόλ Γκάλος από τον σύλλογο των δικηγορικών του Βελγίου που θα μας μιλήσει για τα προβλήματα που αντιμετώπισαν οι δικηγόροι που ασχολούνται με αυτό το ζήτημα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όταν ε, αναλύουμε την ομολογία το Βέλγιο για θέματα απαγωγών τέκνων μπορούμε να δούμε ότι υπάρχουν τέσσερις βασικές δυσκολίε. Αναφέρομαι στην πρώτη διότι δεν αφορά τα ε, κράτη της Ένωσης αλλά τα τρίτα κράτη. Πρόκειται για την σόρευση των εφαρμοζόμενων συμβάσεων, Χάγης, Λουξεμβούργου κλπ. Αυτό δεν μας αφορά. Η δεύτερη δυσκολία ανάγεται στον ορισμό του συνήθου τόπου διαμονή του τέκνου. Ε, τα δικαστήρια αναφέρονται συχνά σε έναν ορισμό ο οποίος έχει γίνει από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αλλά μερικές φορές είναι δύσκολο να εφαρμοστεί και να ερμηνευθεί δεδομένων των ε, στοιχείων που πρέπει να ληφθούν υπόψη που για να προσδιοριστεί αυτός ο όρος της συνήθους διαμονής. Η δυσκολία αφορά την παράνομη ε, μετακίνηση ε, σύμφωνα με την έννοια της ε, επιμέλειας. Ε, γνωρίζουμε την γονική μέρημνα, γνωρίζουμε την προστασία κλπ. Αλλά αυτό την γνωρισμό δεν τον γνωρίζουμε στο δικαίωμα μας. Και τέταρτο, η βασική δυσκολία αφορά την εφαρμογή των εξαιρέσεων στον γενικό κανόνα της άμεσης επιστροφής του τέκνου η οποία βασίζεται στο ε, τεκμήριο της ε, επιστροφής λόγω του συμφέροντος του τέκνου και εδώ το συμφέρον του τέκνου γίνεται αντιληπτό με τρόπο ε, απροσδιόριστο και πάλι στο όνομα του συμφέροντος του παιδιού αυτό το τεκμήριο συμβατότητας με την άμεση επιστροφή γνωρίζει εξαιρέσεις, εξαιρέσεις ε, αφορούν το σοβαρό κίνδυνο ή τον κίνδυνο τον οποίο διατρέχει το τέκνο. Αυτές οι εξαιρέσεις λοιπόν προβλέπουν συγκεκριμένη εξέταση του τέκνου, δηλαδή μια, ανάκριστα λέγαμε, του τέκνου, ε, με εξέταση λοιπόν, η οποία είναι το σου το μάλλον απαραίτητη, λαμβάνοντα υπόψη την εφαρμογή του άρθρου 3 της Συμβάσεως της Νέας Υόρκης για τα δικαιώματα του τέκνου. Όταν λοιπόν θέλουμε να αναλύσουμε το συγκεκριμένο συμφέρον του τέκνου, αναπόφευκτα έχουμε μια παράταση των διαδικασιών, διότι πρέπει να αναλύσουμε συγκεκριμένες καταστάσεις, υπάρχει προβληματική τη ακρόαση του τέκνου, υπάρχει προβληματική των ε, διαφόρων μέσων προσφυγής και όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα την επιμήκυνση του χρονικού διαστήματος και αυτό ε, παγιώνει κάποιες καταστάσεις, ε, το τέκνο ε, θα γίνει αντιληπτό ως κάτι το δύσκολο και ότι το παιδί ενδεχόμενα να υποστεί κάποιες συνέπειες σοβαρές τώρα. Υπάρχουν εμπόδια τον Γενικό Κανόνα για την άμεση επιστροφή. Πρώτη, ε, πρώτο εμπόδιο είναι η διαδικασία και το δεύτερο αφορά σε αυτήν την ε, σύγκρουση ανάμεσα στο συμφέρον του παιδιού ως κοινό κανόνας αφηρημένος και το συμφέρον του παιδιού που γίνεται αντιληπτό ως συγκεκριμένο συμφέρον που προσδιορίζεται βάσει συγκεκριμένων καταστάσεων και συνθήκων. Το πέρασμα του χρόνου λοιπόν θα δημιουργήσει κάποιο χρονικό συστατικό και έτσι και αυτό είναι που ήθελαν να αποκλείσουν οι Βρυξέλλες 2 και η Σύμβαση της Χάγης. Είχα προετοιμάσει κάποια παραδείγματα νομολογίας αλλά επειδή είναι περιορισμένος ο χρόνος μου θα περιοριστώ σε μία περίπτωση που νομίζω πως συνοψίζει αυτά τα οποία βρίσκουμε στην βελγική νομολογία πρόκειται μια απόφαση του Δικαστηρίου των Βρυξελών της 11 Φεβρουαρίου 2010. Το δικαστήριο αποφαίνεται το 2010 ενώ η ε, παράνομη μετακίνηση είχε, ε, είχε γίνει το Απρίλιο 2008, δύο χρόνια νωρίτερα και το δικαστήριο ε, αρνείται να επιβάλλει την μετακίνηση του τέκνου, την επιστροφή του τέκνου και όταν ε, το φάκελος δεν εξετάζεται άμεσα τότε το... η θέση στην οποία βασίζεται η άμεση επιστροφή δηλαδή η μετακίνηση υπέρ προς την ε, συνήθη προς συνήθι τόπο ε, δια, τότε δεν υλοποιείται και το τέκνο είναι πολύ εγκύτερα στην, ε, στο νέο πλαίσιο ε, ζωής το οποίο δημιουργήθηκε στο, τα δύο εφτά χρόνια. Και το δικαστήριο λέει ότι η επιστροφή του τέκνου δεν μπορεί να εντέλεται αυτόματα ή με μηχανικό τρόπο, ε, εξαρτάται από ειδικέ ατομικές προσωπικές περιστάσεις και θα πρέπει να εκτιμάται κατά περίπτωση. Κάτι το οποίο ε, επιβάλλει να γίνει μια ανάλυση που διαρκεί κάποιο χρονικό διάστημα. Ε, αυτός ο κανόνα λοιπόν της άμεσης επιστροφής ε, σύμφωνα με το συμφέρον του τέκνου και αυτό δεν εμποδίζεται ε, από ένα χρονικό διάστημα. Έχουμε δύο απόψεις. Πρώτη αφορά στην έννοια του συμφέροντος του τέκνου και τον ε, λειτουργία που διαδραματίζει αυτό. Όταν διαβάζουμε λοιπόν τις αποφάσεις του δικαστηρίου της ε, Νέας Υόρκης διαπιστώνουμε ότι το συμφέρον του τέκνου μπορεί να μην έχει τη λειτουργία είτε πρόκειται για θέματα διαδικασίας είτε για θέματα ουσίας και αυτή είναι μια διαφορά που θα μπορούσε να ε, ληφθεί υπόψη ότι, το, ότι η έννοια του συμφέροντος του παιδιού μπορεί να μην είναι η ίδια ε, αν, ανάλογα εάν εξετάζουμε το θέμα από ποια πλευρά μάλλον εξετάζουμε το ζήτημα Ο ε, δεύτερος τρόπος είναι να αναθεωρήσουμε τη διαδικασία όπως προβλέπετε από τον κανονισμό Βρυξέλλες 2α δεν θα επανέλθω στα όσα ήδη ελέγχθησαν αναφορικά με την μεταρρύθμιση αυτή. Υπάρχουν δύο άξονες. Ο πρώτος είναι να τονίσουμε το θέμα της διαμεσολάβησης. Νομίζω πως οι όλοι οι επαγγελματίε γνωρίζουν ότι η δικαστική διαδικασία δεν είναι απαραίτητο προσαρμοσμένη στο θέματα ε, οικογενειακού δικαίου και είναι ακόμα πιο επίγον εάν υπάρχει μια κατάσταση που θα πρέπει να αποκατασταθεί έτσι ώστε να αποφευθεί κάθε ρήξη των οικογενειακών σχέσεων που πρέπει να προωθήσουμε την διαμεσολάβηση, όχι μόνο να την οργανώσουμε, αλλά να την προωθήσουμε και να ενημερώσουμε το κοινό, να το παροτρύνουμε για την υλοποίηση. Όταν δεν είναι δυνατόν λοιπόν και βρισκόμαστε στο πλαίσιο δικαστικής ε, ε, διαμάχες, τότε θα πρέπει να καθορίσουμε κάποιο ε, ημερολόγιο, κάποιο χρονοδιάγραμμα, σύμφωνο με, την, ε, με τον κατεπίγοντα χαρακτήρα της υπόθεσης, δηλαδή η μείωση του αριθμού των προσφυγών, άρα εξειδικευμένοι δικαστές για θέματα απαγωγής, σημαίνει επίσης ε, ύπαρξη ε, ποινών σε περίπτωση μη επιστροφής του τέχνη και αναφέρθηκε επίσης στο ζήτημα της ε, διαδικασίας ex equator. Σήμερα υπάρχει η δυνατότητα επιστροφής σύμφωνα με το πλαίσιο 11.6, αλλά την τελευταία λέξη την έχει το κράτος καταγωγής που μπορεί να ακολουθεί τη διαδικασία χωρίς την ε, κήρυξη εκτελεστότητας. Διαφορετικά θα αντιμετωπίζουμε καταστάσει ιδιαίτερα περίπλοκε. Ε, σκεφτείτε μία απόφαση επιστροφής που λαμβάνεται σε ένα κράτος ε, καταφύγιο οι γονείς ε, που έχουν απαγάγει το παιδί ε, ε, πηγαίνουν σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα και θα πρέπει να ακολουθήσουν ή τη διαδικασία μετά ex equator ή την κήρυξη εκτελεστότητας ή να ακολουθήσουν αυτή που προβλέπει το κράτος στο οποίο έχουν καταφύγει. Θα ήταν χρήσιμο επίσης να ξανασκεφτούμε αυτή τη διαδικασία του άρθρου 11.6, δηλαδή ότι την τελευταία λέξη την έχει το κράτος ε, καταγωγής, όταν αυτό το κράτος εκδώσει ε, απόφαση επιστροφής, αλλά πρέπει να τηρήσει κάποιες προϋποθέσεις και ειδικά την ακρόαση του τέκνου, εκτός αν το τέκνο έχει τέτοια ηλικία που ε, δεν καθίστερε δυνατή μια παρόμοια ακρόαση. Κάποιε περιπτώσει λοιπόν μπορεί να υπάρχει πρόβλημα. Γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει ε, ε, ε, εξίσωση αυτών των κανόνων. Και όταν ο γονέας που έχει επαγάγει το παιδί αρνείται να μετακινήσει το τέκνο, να το επιστρέψει, τότε θα πρέπει να περάσει υπόθεση από τα δικαστήρια έτσι ώστε να μπορέσει να εφαρμοστεί η απόφαση. Θα πρέπει λοιπόν το κράτος ε, το οποίο έχει καταφύγει, ο γονέας ε, να προβλέψει μέτρα προστασίας, ε, δηλαδή να υπάρξει αναγνώριση και εκτέλεση στον χώρα καταγωγής του παιδιού. Αυτό μπορεί να συμβάλλει σε κάποιες διαδικασίες συντόμευσης των διαδικασίων. Ευχαριστώ πολύ. Δόκτωρα Γκάλος, τώρα έχουμε τη δυνατότητα ερωτήσεων. Λοιπόν, έχουμε κάποια λεπτά που μας απομένουν. Μπορούμε να προσθέσουμε και άλλα λεπτά. διότι έχουν ξεκινήσει και με καθυστέρηση ερωταπαντήσεις. Yes, Mrs. φαντάστηκα κύριε Ζεύκα, επειδή εσεί είστε συγκητή, θέλετε πρώτο να πάρετε το λόγο. Εν περιπτώσει, θα πρέπει να πω ότι χαίρομαι που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, υπέβαλε αυτό το σχέδιο και η δική μου έκθεση την οποία συνέταξα τον Νοέμβριο του 2016 την έψαξα και διαπίστωσα ότι ορισμένε από τις προτάσεις που είχα τότε διατυπώσει εγώ πραγματικά αντανακλώνται στην πρόταση της Επιτροπής και βεβαίως αυτό για μένα είναι θαυμάσιο. Και ε, εδώ με αυτό εννοώ και ένα, ε, την προτεραιότητα που δίδεται στο, στη διαμεσολάβηση ε, όλες αυτές οι εμπειρίες της, ε, του γαλλογερμανικού μοντέλου που εκπονήθηκε τότε ε, φαίνεται ότι ε, γίνονται αποδεκτές. Εδώ γύρεται το εξή θέμα. Θα πρέπει οι προθεσμίες να είναι σύντομες. Από την άλλη θέλουμε να γίνεται σωστά η διαμεσολάβηση, άρα χρειάζεται κάποιος χρόνος. Και βεβαίως θα πρέπει να εξασφαλίσουμε όταν οι γονείς αποτέχονται μια διαμεσολάβηση, κάτι το οποίο βεβαίως δεν είναι υποχρεωτικό για αυτούς, τότε ε, θα πρέπει να υπάρχει, ε, να συμπεριληφθεί και το ζήτημα της παραγραφής. Θεωρώ ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό για να μην ε, γίνεται κατάχρηση αυτής της διαδικασίας προκειμένου να δημιουργείται ένα τελεσμένο εδώ. Θεωρώ ότι αυτό είναι το, αυτό είναι σημαντικό αυτό το θέμα. Είπατε ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με τον χειρισμό των ενιών. Ε, γι' αυτό και εμείς δεν μιλάμε για απαγωγή entführung ε, στα γερμανικά αλλά για entziehung ε, απομάκρυνση του παιδιού. Ε, το, το οποίο σημαίνει ότι ο ένας γονέας ε, αρπάζει το παιδί και φεύγει ε, ε, χωρίς να έχει συνείδηση ότι κάνει κάτι παράνομο. Δεν πρόκειται για απαγωγή εδώ, πρόκειται για αφαίρεση, απομάκρυνση του παιδιού, ε, φαινόμενο στο οποίο, το οποίο δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζει με τέτοια αυστηρότητα ο νόμος όπως μια υπόθεση απαγωγής. Νομίζω ότι πρέπει αυτό κάπως να το λάβουμε υπόψη και να το διαφοροποιήσουμε. Ε, χαίρομαι πολύ για την ε, μελλοντική ε, επεξεργασία όλων αυτών των θεμάτων και θεωρώ ότι πραγματικά έχουν συμπεριληφθεί πολύ σωστά στοιχεία. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Κέπχαρτ. Ο κύριος Τζέφκα. Ταντεουζεύκα, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ όλα τα μέλη του πάνελ. Εξαιρετικά ενδιαφέροντα αυτά που είπαν. Ευχαριστώ τους εκπροσώπους και του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτά που υπόθηκαν θεωρώ ότι ήταν πολύ θετικά. Παρόλο που το θέμα της συζητήσεως είναι περιπλοκότατο και άκρος ευαίσθητον. Προχωρούμε. Δεν υπάρχουν φραγμοί από πλευράς κρατών μελών. Και βλέπουμε ότι υπάρχει η ανάγκη να καταλήξουμε σε αποτελεσματικότερα εργαλεία ή να προσαρμόσουμε τα εφιστάμενα. Και σίγουρα αυτό θα παίξει ρόλο στις διαπραγματεύσεις μας. Και ελπίζω να καταλήξουμε σε ένα αίσιο τέλος. Παρ' όλα αυτά έχω την εντύπωση όποτε αναφέρομαι στο ενδιαφέρον αυτό ζήτημα και όποτε ακούω κάποιους να εκφράζουν την άποψή τους γι' αυτό, ότι εν γέννη επαναλαμβάνουμε ότι το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού είναι η βασική μας μέρημνα. Και αυτός είναι ο λόγος που ψάχνουμε κάποιες νομικές λύσεις. Πίσω από αυτό πάντα βρίσκεται και το συμφέρον του γονέα. Υπάρχει σχέση λοιπόν μεταξύ συμφερόντων του παιδιού, του γονιού, του ενήλικα, του κράτους μέλους. Υπάρχουν διάφορα αλληλένδα συμφέροντα. Εξού και ερώτησή μου οι φόβοι που δημιουργούνται και δημιουργήθηκαν στο Συμβούλιο όταν συζητούσαμε εκεί το θέμα. Για να απαλλαγούμε από τη διαδικασία της, του εκτελεστού, όταν απαλλαγούμε από το εξεκουάτορ, θα μειωθεί ο αναγκαίος χρόνος για τις διαδικασίες. Και αυτό είναι κρισίμου σημασία για την προστασία των συμφερόντων του παιδιού. Το δεύτερο που θέλω να αναφέρω είναι ότι έχω κάποια εμπειρία και θέλω τη δική σας άποψη όσον αφορά τις ακροάσεις των παιδιών. Είμαι βαθύτατα πεπισμένος ότι η ακρόαση του παιδιού είναι κάτι υποχρεωτικό. Δεν που δεν είναι αυτό. Όμως θα συζητηθεί το σε ποια ηλικία μπορεί να ακουστεί άποψη του παιδιού σε ποια ηλικία το παιδί μπορεί λογικά να παρουσιάσει μια κατάσταση, μια θέση που μπορεί να είναι αποδεκτή. Πότε μπορεί να εκφράσει την άποψή του ή την άποψή της το παιδί. Το τρίτο θέμα. ποια είναι η υπεύθυνη αρχή που θα αναφέρεται στον κανονισμό. Για κάποιες ε, δεν υπάρχουν οικογενειακά δικαστήρια σε κάποιες χώρες, σε κάποιες υπάρχουν. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περιορίζει τον αριθμό των κεντρικών αρχών του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνε για τα θέματα αυτά, για τον καθορισμό γονικής ευθύνης ή για την απαγωγή των παιδιών. Εγώ θα ακολουθήσω, θα χρησιμοποιήσω αυτή την ορολογία. Απαγωγή παιδιών. Ο γονιός καμιά φορά καταλαβαίνει ότι έχει απαγάγει το παιδί. Αυτά λοιπόν ήθελα να αναφέρω, αυτά τα τρία στοιχεία στον τομέα που συζητούμε. Και αυτά είναι σημεία που με προβληματίζουν και θα ήθελα να τα αναλύσω. Ο κύριος Λιμπρετών. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω όλους που πήραν το λόγο, όσους ήρθαν σήμερα να μιλήσουν για διατύπωση του κανονισμού Βρυξελών 2α. Είναι σημαντικότατο πρόβλημα ανθρώπινο. Είναι θέμα διασυνοριακών οικογενειακών συγκρούσεων. διεθνείς απαγωγές παιδιών. Συζητούμε. Στην εκλογική μου περιφέρεια έρχονται γονείς και με βρίσκουν που θεωρούν ότι είναι θύματα τέτοιων απαγωγών. Δεν ξέρω αν είναι κάτι ιδιαίτερο και ειδικό. Πολλή φορά, πολλές φορές είναι ε, παιδιά ε, Γάλλοι που απάγονται. Δεν ξέρω αν αυτά τα συχνά φαινόμενα συμβαίνουν μόνο στην εκλογική μου περιφέρεια και κύμα Ήδη ήξερα με υπόθεση διαμεσολάβηση Γάλλο-Γερμανική παλιά. Νομίζω ότι είναι διαδεδομένο το φαινόμενο. Πρέπει να βρεθούν λύσει. Αναφέρατε κάποιε λύσει. Μέσω διεθνού οικογενειακή διαμεσολαβήσεω. Ενδιαφέρθηκα από την παρουσίαση εκείνου που εκπροσωπούσε τον οργανισμό ΜΙΚ. Έχω ένα στόχο που ευχάριστο με εξέπληξε. 65% των διαμεσολαβήσεων ΜΙΚ καταλήγουν σε συμφωνία. Κατάλαβα σωστά. Εάν έτσι έχουν τα πράγματα, αυτό είναι ένα παράδειγμα προς πρόθεση και προς έμπνευση. Το άλλο που με ενδιαφέρει. Η καλύτερη συνεργασία μεταξύ κεντρικών αρχών. Σωστά τα κατάλαβα. Δηλαδή πρέπει να πείσουμε να δημιουργηθούν ειδικά μαθήματα για την κατάρτιση που αφορούν σε Αυτό θα επέλυε το πρόβλημα. Το τελευταίο πρόβλημα. Η κατάργηση της εντολής εκτελεστού. Πολλοί το ανέφεραν αυτό. Εγώ έχω αμφιβολίες. Δεν είμαι τόσο ενθουσιώδης γι' αυτό. Μίσος έτσι πλήττεται η κυριαρχία των κρατών και μάλιστα κατά υπερβολικό τρόπο. Αυτά προς σκέψη. Ευχαριστώ κύριε Λεμπρετών. Κάποιες ερωτήσεις ετέθησαν. Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ξεκινήσει. Δόκτωρ Πάολ, να γίνει κάποια προσπάθεια απάντησης. Να μην απαντούν όλοι σε όλες τις ερωτήσεις σας παρακαλώ όμως. Δόκτωρ Πάολ, ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να απαντήσω στις τεθείς ερωτήσεις. Καταρχήν θα μιλήσω γερμανικά γιατί βάζω ε, την ερώτηση στα γερμανικά. Αναφερθήκατε στην ανάγκη να τηρούνται προθεσμίες και πραγματικά έχετε δίκιο. Αυτή είναι μια από τις μεγαλύτερες δυσκολίες όταν βλέπουμε πόσο απίστευτες είναι οι συγκρούσεις που φέρνουν οι γονείς σε τέτοιου Η διαμεσολάβηση είναι μια διορθωμένη διαδικασία και βεβαίως ε, θα πρέπει να συμπυκνώσει κανείς αυτή την δομή της διαμεσολάβησης, να τη συρρυκνώσει ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και αυτό είναι πολύ δύσκολο, εάν θέλει βεβαίως παράλληλα να λάβει υπόψη της ε, ανάγκης, ε, της τις των γονέων αυτούς που απάγουν, ε, το παιδί, αυτούς που μένουν πίσω κλπ. Ε, είναι δύσκολο, είναι τη διαδικασία. Παρ' όλα αυτά ε, πετυχαίνει αρκετά συχνά όταν είναι επαρκής η εκπαίδευση των διαμεσολαβητών. Εμείς η υπόθεση εκδικάζεται ενώπιον του δικαστηρίου. Ε, και στη συνέχεια γίνεται η διαμεσολάβηση επί δύο ή τρεις, ε, για δύο ή τρεις μέρες. Όσον αφορά τον αριθμό των υποθέσεων και το ποσοστό επιτυχίας, δεν είναι 75-65%. Τώρα μιλήσατε για τις ιδιαιτερότητες των γαλλογερμανικών σχέσεων. Η Γερμανία έχει τα περισσότερα γειτονικά κράτη στην Ευρώπη, περισσότερα σύνορα και έχουμε τον ίδιο αριθμό συγκρούσεων με τους Γάλλους, με τους Πολωνούς, με τους Ολλανδούς, με τους Ελβετούς, τους Αυστριακούς. Άρα είναι τυπικό πρόβλημα και των γειτονικών χωρών μας. Η πρωτοβουλία του γαλλογερμανικού σχεδίου ήταν πρωτοβουλία των Γάλλων και των ε, Γερμανών, των Υπουργών Δικαιοσύνης Είπαμε εμεί σαν εταίροι ότι είχαμε, περνάγαμε δύσκολες περιόδους ιστορικά και να έπρεπε να δοκιμάσουμε κάτι καινούριο. Αυτό ήταν κάτι ιδιαίτερο και η κυρία Γκέπχαρτ θα σας το επαναλάβει αυτό πιστεύω. Ρωτάτε πώς τα πάμε, πώς καταφέρνουμε να πετυχαίνουμε το 65%. Δεν είναι εύκολο. Πολλές τέτοιες υποθέσεις έχω εξετάσει και έχω ασχοληθεί. Δεν πέτυχαν όλους. Όταν τα... υπάρχει μια καλή προετοιμασία, εμείς έχουμε το ΜΙΚ, όταν υπάρχει υπηρεσία καλή που προετοιμάζει τη μεσολάβηση, προετοιμάζει τα μέρη για τη διαδικασία διαμεσολάβησης, ενθαρρύνει τα μέρη για διαμεσολάβηση και υπάρχει καλή συνεργασία με τους δικαστές και τις κεντρικές ε, αρχές και υπάρχει και ευλογία του δικαστηρίου του ΣΥΠΗΝ, τότε τα μέρη είναι τόσο ικανοποιημένα και τόσο ευγνώμονα που ε, τους δίδετε χρόνο και τους βοηθάτε που πετυχαίνουμε. Με σκληρή δουλειά τα καταφέρνουμε. Αυτή είναι η απάντηση. Σκληρή δουλειά. Ευχαριστώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. πάνω σε αυτά που μας είπε ο Δόκτωρ Πολ. Πράγματι, η δημοσιολάβηση χρειάζεται χρόνο. Και είναι ήδη μια σύντομη διαδικασία. Υπάρχουν πολλές καλές πρακτικές. Το ΜΙΚ είναι μία από αυτές. Στο Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο προσπαθούμε να ανταλλάξουμε βέλτιστες πρακτικές. Και βλέπουμε πώς εντάσσεται η διαδικασία διαμεσολάβηση. Όπως στην Ολλανδία. Όταν γίνεται αυτό λειτουργεί άριστα και είναι επιτυχέστατη ακόμα και σε σύντομο χρονικό διάστημα είναι δυνατόν να ολοκληρωθούν διαδικασίες περί απαγωγής. Για, το, για την παραγραφή δεν θα πρέπει η διαμεσολάβηση να έχει κάποια αρνητική συνέπεια όσον αφορά την παραγραφή. Έχουμε κανόνες, έχουμε την οδηγία διαμεσολάβησης όπου αυτό προβλέπεται. Προβλέπεται όταν τα μέρη έχουν προσφύγει στη διαμεσολάβηση η χρονική περίοδος για την παραγραφή αναστέλλεται κατά τη διάρκεια της διαμεσολάβησης. Η διαμεσολάβηση δεν έχει αρνητικό αντίκτυπο για οδήποτε μέρος που θέλει μετά να διεκδικήσει δικαιώματα στο δικαστήριο. Όσον αφορά την ακρόαση του παιδιού, κύριε Τζέφκα, είπατε ότι ιδεοδός θα πρέπει να έχουμε κοινά πρότυπα και προδιαγραφές, αυτό θα ήταν το ιδεώδες. Το συζητήσαμε ενδελεχέστατα στην ομάδα εμπειρογνωμόνων το θέμα αυτό. Νομίζουμε ότι οι πρακτικές ποικίλουν ευρέως στα κράτη-μέλη και οι απόψεις και οι νοτροπίες όσον αφορά την ακρόση του παιδιού ποικίλουν και θα ήταν συνεπώς δυσχερέστατο να καταλήξουμε σε κοινή αντίληψη όσον αφορά την ηλικία που αποτελεί όριο για, το, για την ακρόση του παιδιού και είναι κάτι ευμετάβλητο η ηλικία Κάποια παιδιά ρημάζουν πιο γρήγορα από άλλα. Η ηλικία, πώς να γίνει ακρός του παιδιού. Το να καταλήξουμε σε κοινή αντίληψη για αυτές τις πρακτικές θεωρούμε ότι είναι κάτι αρκετά δύσκολο. Ενώ αμοιβαία αναγνώριση των συστημάτων μας είναι κάτι πιο εφικτό και επαρκές που θα εξασφάλιζε την ελεύθερη κυκλοφορία των αποφάσεων. Ετέθηκε θέμα και για την εντολή εκτελεστού, εκτελεστότητα στην Ευρώπη ξεπεράσαμε το θέμα της κυριαρχίας. Αυτός ο κανονισμός ήταν ο πρώτος στον οποίο το εξεκουάτορ καταργήθηκε για κάποια δικαιώματα και εντάλματα επιστροφής ήταν κάτι που έδειξε την πολιτική βούληση να κινηθούμε προς σωστή κατεύθυνση. Και μετά στον τομέα της δικαιοσύνης γενικότερα συνεχίσαμε σε θέματα μικρών ισχυρισμών, διατροφής κλπ εμπορικές αξιώσεις στα πλαίσια του κανονισμού Βρυξέλλες 1. Άρα είμαστε έτοιμοι να επεκτείνουμε την ίδια προσέγγιση και εδώ. Αυτές τις ερωτήσεις σημείωσα, ίσως να υπάρχουν και άλλες, αλλά και άλλοι θα έχουν άλλα να πούν. Εσείς, ευχαριστώ για τις ερωτήσεις, διότι δεν είχα πρόθεση να πω ότι θα πρέπει να αλλάξει το όνομα. Πρέπει να κάνουμε διακρίσεις στις περιπτώσεις. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου μπορούμε να μιλούμε για απαγωγή, για αφαίρεση, αρπαγή κλπ. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις όπου η παράνομη ή νόμιμη μεταφορά είναι πάρα πολύ λεπτή η μετακίνηση διότι εξαρτάται από αυτήν η νομιμότητα της, η, η, παρανομία της μετακίνησης ε, αφορά αυτό που λέει και στην του Βέλγιο. Το δικαίωμα του γονέα να μεταφέρει τον τόπο διαμονής ε, του παιδιού ε, είναι δυνατόν, αλλά νομίζω ότι δεν μπορούμε να συγκρίνουμε περιπτώσεις που είναι στα όρια της νομιμότητας σε σχέση με την κυριότητα θα έλεγα του τέκνου και να αποκλείσουμε την ε, σχέση με τον άλλο γονέα. Να γίνει αυτή η ρήξη της σχέσης. Οι, οι δύο αυτές περιπτώσεις, ε, εάν τις ε, συγκρίνουμε, μάλλον όπως έχουν τώρα, θα πρέπει να ξαναπαθεωρηθούν. Τώρα, ο ο δικαστής και τα, τα δικαστήρια είναι ένας τρόπος για να δώσουμε να γίνει κατανοητός σε όλους και σε όλα τα κράτη τι είναι προς το συμφέρον του παιδιού. Ε, λοιπόν, εάν λοιπόν αυτή η γοργή και η άμεση επιστροφή θα πρέπει να γίνει πάση θυσία ή θα πρέπει να σταθμίσουμε τις περιπτώσεις. Αυτό μπορεί να γίνει ε, μόνο αν έχουμε συγκεκριμένους δικαστές, επαγγελματίες που θα αναλαμβάνουν και θα επιλαμβάνουν αυτών των καταστάσεων. Αυτό νομίζω είναι ιδιαίτερα σημαντικό και επανέρχομαι τώρα στο ζήτημα της ακρόασης ε, του τέκνου που έθεσε ο κύριος Βουλευτής διότι η ακρόαση του τέκνου είναι ένα ζήτημα πολύ λεπτό διότι όλοι γνωρίζουν πως το τέκνο μπορεί να εκτεθεί σε κάποιες καταστάσεις που έχουν αρνητικές επιπτώσεις στον γονέα που δεν θα επιλεγεί. Είναι λοιπόν ένας χώρος στον μπορεί να ε, παρέμβει η διαμεσολάβηση γύρω από το θέμα της ακρόασης και της τήρησης της αξιοπρέπειας του τέκνου και ειδικά για να μην δώσουμε στα, στο παιδί ε, τη βαρύτητα της απόφασης δεν είναι δηλαδή όλο όλο αδιάφορο αυτό. Πρέπει να υπάρχουν κάποια πρότυπα παραδεκτά, όχι ενοποιημένα, ενία αλλά δεν θα πρέπει να ζητήσουμε από το παιδί να απαντήσει με ποιον γονεί επιθυμείς να παραμείνεις. Αυτά είναι σημεία τα οποία ήθελα να τονίσω. Η Δόκτωρ Γκάλλας. Να προσθέσω κάτι σχετικά με την ακρόαση του τέκνου. Συμφωνώ με τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να είναι αυτή η ομοιογένεια. Θα πρέπει να ε, γνωρίζουμε το ζήτημα ε, ε, ε, λάβουμε υπόψη. Μήπως μπορείτε να μιλάτε λίγο πιο αργά παρατηρεί ο Πρόεδρος. Έλεγα λοιπόν προς το συμφέρον του τέκνου να έχουμε έναν ενιαίο κανόνα για, τις, τον τρόπο που θα εξεχθεί η ακρόαση. Θα είναι πολύ περίπλοκο διότι αυτή, υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση που ανάμεσα στα κράτη-μέλη για το θέμα της ηλικία και τώρα για τον κύριο Λεμπρά να πω ότι αυτά τα δύο πράγματα που αναφέρατε είναι συμπληρωματικά. Αυτό ε, η ιδέα της εξειδίκευσης ε, ε, υπάρχει. Έχουμε μόνο πέντε δικαστήρια για οικογενειακά ζητήματα όπου υπάρχει και ένα εφετείο και αυτά τα πέντε δικαστήρια θα πρέπει και να εξετάσουν αυτές τις παράνομες μετακινήσεις. Δηλαδή πέντε δικαστήρια τα οποία έχουν εξειδικευτεί με ε, δικαστές που συνδιαλέγονται μεταξύ τους έτσι ώστε να μπορούν να οδηγηθούν σε μια ενιαία κατά κάποιο τρόπο απάντηση για αυτές τις περιπτώσεις απαγωγής. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων. Προτείνω να περάσουμε στο δεύτερο πάνελ μας που αφορά στη συνεργασία ανάμεσα στις κεντρικές και δικαστικές αρχές για τον λόγο φυσικά της αναδιατύπωσης της, ε, του κανονισμού και θα ήθελα να εστιάσετε στο θέμα της ε, ε, διασυνοριακής συνεργασίας και να ακούσουμε κάποιες εμπειρίες από κάποιες κεντρικές αρχές στην Τσεχία και έναν ανώτατο δικαστικό από τις κάτω χώρες, ο Δ από το Πανεπιστήμιο της Αμβέρσας. Παρακαλείτε να λάβει το λόγο για 10 λεπτά. Ευχαριστώ. Thank you very much. Good afternoon. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σε όλους. Σας ευχαριστώ πολύ που μου δώσετε την ευκαιρία να παρίσταμε εδώ σήμερα. Μου ζητήθηκε να μιλήσω για την ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας. Αυτό το οποίο διαπιστώσαμε είναι ότι η Κομισιόν έκανε ήδη πολλά στην κατεύθυνση αυτή. Νομίζω ότι υπάρχουν πολλές καλές προτάσεις και αυτό το οποίο έκανα εγώ στις μου διαφάνειες είναι να βάλουμε επιχαίως ε, γράμματα αυτά τα οποία ήδη έκανε τα... που έκανε ήδη η Επιτροπή και στη συνέχεια αυτά που μπορεί να, που μπορεί να επιφέρει το Κοινοβούλιο. Καταρχήν η διάρκεια των ε, υποθέσεων. Ε, η Επιτροπή είπε ότι οι κεντρικές αρχές θα πρέπει να ανταποκρίνονται στα αιτήματα εντός δύο μηνών. Είναι πολύ καλό να βάλουμε μια χρονική προθεσμία, ωστόσο θεωρώ ότι θα υπάρξουν περιπτώσεις που είναι πιο επίγουσες, γιατί η διάρκεια αυτή είναι υπερβολικά μεγάλη ε, και δεν θα πρέπει να υπάρξει να λειτουργήσει σαν δικαιολογία για να διαρκέσει η διαδικασία αυτή δύο μήνες. Όταν είναι επίγουσα λοιπόν η ετούσα κεντρική αρχή θα πρέπει να ζητήσει από την άλλη αρχή στην οποία να απευθύνει το αίτημα να ανταποκριθεί σε μια βραχύτερη περίοδο. Ε, στην πρόταση της Επιτροπής ε, αναφέρεται η διάρκεια των έξι εβδομάδων. όσον αφορά την ε, διοίκηση, δηλαδή την κεντρική αρχή και την ακροματική διαδικασία στο δικαστήριο. Νομίζω ότι είναι πολύ καλή αυτή η διευκρίνηση και θα μπορούσαμε να διευκρινίσουμε περαιτέρω ότι το άρθρο αυτό αναφέρεται στη περίοδο μέχρι την εμφάνιση στο δικαστήριο ή την υποβολή στο δικαστήριο. Το δεύτερο είναι το θέμα του κόστους κάθε κεντρική αρχή θα πρέπει να υπολογίσει το, τις δικές της δαπάνες, αλλά θα πρέπει να υπάρξει μια ευελιξία ε, στην περίπτωση για παράδειγμα που θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία με άλλες αρχές ώστε μπορεί να γίνει ένας επιμερισμός των δαπανών. Τώρα, όσον αφορά τους δικαστές, ε, ε, οι δικαστές και οι κεντρικές αρχές θα πρέπει επίσης να συνεργάζονται, θα πρέπει αυτό να συμπεριφθεί στην, κεντρική, ιδεολογική σκέψη, θα πρέπει και οι δικαστές να είναι ανοιχτοί σε αυτή τη μορφή συνεργασίας, θα αναφερθώ σε αυτό αργότερα, και θα πρέπει ε, να έχουν και την, το χρονικό περιθώριο οι δικαστές να ανταποκριθούν. θα πρέπει και αυτοί να έχουν ένα χώρο, ε, τη δυνατότητα σχέση με το δικό του χώρο εργασία να ανταποκριθούν. Οι άλλε διαφάνειες αφορούν την ενίσχυση προσωρινών μέτρων και την ενίσχυση των διαταγμάτων επιστροφής του παιδιού, των επιστροφής του παιδιού, ε, που θα πρέπει να είναι άμεσα εκτελεστές. Τώρα, αυτό το οποίο μπορεί να συμβεί είναι ότι μπορεί να έχουμε ένα προσωρινό μέτρο ασφαλιστικό μέτρο το οποίο να ληφθεί στην Ουγγαρία ενώ η Σλοβακία έχει τη δικαιοδοσία για την εκδίκαση της υπόθεσης αλλά τα ασφαλιστικά μέτρα στην περίπτωση αυτή κατα ωστόσο είναι εκτελεστά από την άλλη. Άρα θα πρέπει να υπάρχει μια επικοινωνία εν σχέση με το πότε θα καταπέσουν αυτά τα μέτρα και θα πρέπει οι κεντρικέ αρχέ να συμφωνήσουν ποια μέτρα είναι εκτελεστά και ποια όχι. Και θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει μια υποχρέωση για τα δικαστήρια να ενημερώνουν την κεντρική αρχή στη χώρα στην οποία έχουν λεφθεί τα ασφαλιστικά μέτρα. Ε, για την περίπτωση που έχουν καταπέσει ούτως ώστε να το γνωρίζουν οι κεντρικές αρχές. Το ίδιο ισχύει και για τα, την εντολή επιστροφής του παιδιού, την απόφαση επιστροφής του παιδιού ε, όσον αφορά μια απόφαση επί της ουσίας. Ε, αν υπάρξει μια άλλη απόφαση επί της ουσίας θα πρέπει και πάλι ε, να υπάρξει μια επικοινωνία μεταξύ των κεντρικών αρχών ούτως ώστε να γνωρίζουν ποια, τελικά, ποια απόφαση τελικά είναι εκτελεστή, θα πρέπει να γίνει εκτελεστή. Ο κανονισμός αυτή τη στιγμή και στην πρόταση είναι το πρώτο δικαστήριο το οποίο, έχει την, το οποίο επιλαμβάνεται της υπόθεσης το οποίο έχει τη δικαιοδοσία. Ε, πρέπει, όπως είπαμε, να υπάρχει μια άμεση επικοινωνία μεταξύ δικαστών. Εάν επιληφθεί ένα δικαστήριο, αλλά αν ε, έχει προηγουμένως επιληφθεί κάποιο άλλο δικαστήριο, θα πρέπει να υπάρξει ε, μια αμοιβαία ενημέρωση ε, σε σχέση με την ημερομηνία κατά την οποία ε, το πρώτο, ε, κατά την το δικαστήριο πρώτα λήφθη της υπόθεσης. Και αν το κοινοβούλιο το αποδεχτεί, η υποχρέωση αυτή αμοιβαίας ενημέρωσης θα πρέπει να συμπεριληφθεί στις υποχρεώσεις των κεντρικών αρχών που εμπίπτουν στο άρθρο 63. Τώρα, ορισμένες φορές θα πρέπει να εφαρμοστεί το οικογενειακό δίκαιο, όλες φορές το οικονομικό δίκαιο και η Επιτροπή ε, θα πρέπει να παράσχει τις σχετικές πληροφορίες και νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρξει το καθήκον των κεντρικών αρχών να ενημερώσει και την Επιτροπή για μια αλλαγή στην ε, ε, νομοθεσία. Τώρα, η αναγνώριση των αποφάσεων και εφαρμογή. Με την κήρυξη εκτελεστότητας νομίζω ότι η κεντρική αρχή θα πρέπει επίσης να είναι υποθετική σε αυτή τη φάση, έστω, έστω και αν δεν υπάρχει αίτημα εκτέλεση ενός μέτρου, η κεντρική αρχή θα πρέπει να είναι σε θέση να υποστηρίξει τη διαδικασία ε, μετακίνησης και τοποθέτησης ε, του παιδιού. Ε, τώρα, η προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού, το ζήτημα της κρόασης του παιδιού, σημαντικό βήμα θα ήταν επίσης να επιφορτιστεί η κεντρική αρχή, να συνδράμει το παιδί, διευκολύνοντας τη χρήση βιντεοδιασκέψεων πλαισιώνοντας έτσι καλύτερα το παιδί και, και επίσης σχέση κανονισμό για τα αποδεκτικά στοιχεία. Δεν είναι σε όλες τις χώρες ίδιες οι αρμόδιες αρχές, αλλά θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα επαφής, ούτως ώστε να μπορούν να στηρίξουν τη διαδικασία κρόσης του παιδιού. Ε, επίσης θα πρέπει να, οι κεντρικές αρχές να συνδράμουν στην την, ε, ε, μετακίνηση, την τοποθέτηση του παιδιού και να υποστηρίξουν αυτούς που έχουν την ευθύνη του παιδιού είτε γονείς είναι αυτοί είτε κάποιο ίδρυμα. Τώρα, υποχρεώσεις ε, για τα δικαστήρια να λάβουν υπόψη το ενδεχόμενο της αμεσολάβησης, θεωρώ ότι είναι θετικό. Ε, νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να γίνεται όχι μόνο σε περιπτώσεις απαγωγών των παιδιών, αλλά σε όλες τις περιπτώσεις που αφορούν την μέρημνα των παιδιών και θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα ειδικό καθήκον των κεντρικών αρχών να υποστηρίζουν τη διαδικασία διαμεσολάβησης ε, προπαρασκευάζοντας ακριβώς αυτή τη ε, διαδικασία και νομίζω ότι θα πρέπει να έχουν την υποχρέωση είτε να επιφορτιστούν με αυτή την αποστολή είτε να συνεργαστούν με κάποιες αρχές οι οποίες είναι επιφορτισμένες με την προπαρασκευή της εν λόγω διαδικασίας. Ευχαριστώ πολύ. Τέλεια ήταν. τηρήσατε το χρόνο που σας διαθέσαμε, υπήρξατε ακριβέστατοι και δεν με ειδοποίησαν ότι μιλάτε πολύ γρήγορα. Ευχαριστώ. Επόμενος. Κύριος Λούκας Φλίντριχς, την Κεντρική Αρχή της Τσεχικής Δημοκρατίας. Κύριε Φρίντριχς, έχετε τώρα το λόγο για ένα δεκάλεπτο. Σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο και εύχομαι σε όλους ε, ένα πολύ καλό απόγευμα και ευχάριστο απόγευμα. Μιλάμε για την τροποποίηση του κανονισμού Βρυξέλλες 2α και θα εκφράσω την άποψη της κεντρικής αρχής της εχικής δημοκρατίας. Ποια είναι τα καθήκοντά μας. Θα μιλήσω για την αλλαγή όσον αφορά τη συνεργασία μεταξύ αρχών και κάποιες υποθέσεις απαγωγής παιδιών και θα προβώ και σε κάποια σχόλια. Και θα αναφέρω και κάποιες εμπειρίες μας. Λοιπόν, ποιος είναι ο ρόλος μας. Ποιος είναι ο ρόλος του φορέα μας. Είμαστε μια κεντρική αρχή. Δεν είναι κάτι που σχετίζεται με τον κανονισμό Βρυξέλλες 2 και τις απαγωγές παιδιών, αλλά αφορά και διασυνοριακές υιοθεσίε και άλλα ζητήματα. Σύμφωνα με το δικό μας δίκαιο της χώρας μου, είμαστε επιφορτισμένοι με κοινωνική και νομική προστασία των παιδιών. Έχουμε παρόμοιες ευθύνες με κοινωνικούς λειτουργούς. Μπορούμε άμεσα να εργαστούμε με τα παιδιά, να έρθουμε σε επαφή με τα παιδιά, κυρίως σε δικαστικές υποθέσεις που σχετίζονται με τα παιδιά και που εμπεριέχουν διασυνοριακό στοιχείο. Άμεσα λοιπόν μπορούμε να συμμετέχουμε στις ε, διαδικασίες τις δικαστικές, να ακούμε τα παιδιά, να προβαίνουμε σε συνεντεύξεις τα παιδιά, να πηγαίνουμε στο δικαστήριο και να παρακολουθούμε την δικαστική υπόθεση από την αρχή μέχρι τέλους. Και μπορούμε να αντλήσουμε από τις εμπειρίες μας ως κεντρικός φορέας. Και είμαστε ενεργοί και δραστήριοι στη διεθνή προστασία των παιδιών και χάρη σε όλα αυτά είχαμε τη δυνατότητα να ασχοληθούμε και με τη διαμεσολάβηση και να προβούμε και σε ε, κατάρτιση για τη διαμεσολάβηση. Έχουμε προγράμματα που χρησιμοποιούν τις βέλτιστες πρακτικές όπως το μοντέλο Κοχένσκι από τη Γερμανία και από αλλού Έχουμε και ένα σχέδιο για να βελτιώσουμε τα συμμετοχικά δικαιώματα των παιδιών στις εργασίες μας. Και τώρα επιτρέψτε μου άμεσα να αναφερθώ σε διάφορα σημεία του κανονισμού. Βασικά μπορούμε να εντοπίσουμε δύο σημαντικά προβλήματα. Αν η ταχύτητα και η αποδοτικότητα της συνεργασίας μεταξύ κεντρικών αρχών είναι καλή ή όχι. Πολύ συχνά έχουμε καθυστερήσει στην επεξεργασία αιτήσεων. Καμιά φορά χρειάζεται μεγάλο χρονικό διάστημα. Όταν θέλουμε να βρούμε πληροφορίες για ένα παιδί, επί παραδείγματι, κάποιες κεντρικές αρχές διεκπεραιώνουν το αίτημα σε μερικές εβδομάδες ή ένα μήνα, άλλες αρχές μπορεί να χρειαστούν και ένα εξάμεινο ή και ένα χρόνο ακόμα για κάτι τέτοιο. Υπάρχουν διαφορές λοιπόν όσον αφορά τις διάφορες χώρες. Επίσης, υπάρχει και ένα ευρύ φάσμα προσφερωμένων υπηρεσιών και δραστηριοτήτων των κεντρικών αρχών. Τα πρότυπα διαφέρουν από χώρα σε χώρα, όπως ήδη ανέφερα, και αυτό πόρο απέχει από το τέλειον. Θα έπρεπε να έχουμε τους ίδιους κανόνες για όλες τις κεντρικές αρχές. Όμως, κάποιοι κανόνες δεν εκφράζονται σαφώς στον ισχύοντα κανονισμό. Καμιά φορά επίσης οι κανόνες δεν εφαρμόζονται ομοιόμορφα ή με σαφή τρόπο. Αυτό το είπαν άλλωστε και κάποιοι συνάδελφοι εδώ. Το άρθρο 56 πει Όταν πήγαινε ένα παιδί σε ένα άλλο κάτω μέλος, βρίσκεται σε άλλο κάτω μέλος. Τώρα όσον αφορά την πρόταση είναι αρκετά ευαίσθητη η προσέγγιση που ακολουθείτε. Θα μπορούσε να βελτιώσει το χρόνο που απαιτείται, διότι τίθενται κάποιες προθεσμίες. Εν συγκρίση με άλλους κανονισμούς, νομίζω ότι αυτός ο κανονισμός απέδειξε ότι είναι πολύ χρήσιμος στην πράξη. Αυτό που είναι εξίσου σημαντικό είναι να εξασφαλίσουμε επαρκή χρηματοδότηση, οικονομικούς πόρους, για τις εμπλεκόμενες αρχές. Διότι όταν μια κεντρική αρχή έχει ήδη ένα ή δύο ανθρώπους που ασχολούνται με τα πάντα που αφορούν τον κανονισμό Βρυξέλλες 2, πολύ συχνά δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν υποθέσεις απαγωγής εγκαίρως και η ποιότητα των προσπαθειών δεν είναι επαρκής. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να αντιμετωπιστεί. Πρέπει να υπάρχει πολύ καλή στελέχωση και πολύ καλή χρηματοδότηση. Δεύτερον, δεύτερος τομέας. Είναι πολύ καλό που η πρόταση συγκεκριμένα αναφέρει αρμοδιότητες και υποχρεώσεις των κεντρικών αρχών, διότι κατά το παρελθόν η ερμηνεία ποικίλε, ποικίλε σε μεγάλο βαθμό από χώρα σε χώρα. Τώρα όμως στην παρούσα πρόταση για αναδιατύπωση μπορούμε να θέσουμε σαν στόχο ένα βαθμό εναρμονίσεως. Επίσης αναφέρονται οι συνθήκες υπό τις οποίες μπορεί κανείς να ζητήσει παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών όσον αφορά τη γονική ευθύνη κλπ. Άρα οι συνθήκες είναι πολύ σαφέστερες σε αυτό το κείμενο προτείνεται. Να πω μερικά λόγια για την απαγωγή, για τις απαγωγές παιδιών και συναφή ζητήματα. Ο πρώτος προβληματικός τομέας είναι πώς θα τηρούνται οι προθεσμίες. Έχουμε καθορίσει πρόσφατα αυτές τις προθεσμίες, διότι μέχρι τώρα Παρόλο που οι κεντρικές αρχές υποτίθεται ότι θα κινούνται με τον ταχύτερο δυνατό τρόπο, αυτό δεν ίσχυε πάντα. Δεύτερο ζήτημα, ο μηχανισμός επιστροφής, αυτός καθεαυτός, ο οποίος θα πρέπει να συνδέεται σωστά με τις εκδικάς των υποθέσεων στα κράτη-μέλη. Άρα χρειαζόμαστε εξειδικευμένα δικαστήρια. Αυτό που ανέφεραν άλλωστε και κάποιοι συνάδελφοι. Επόμενο σημείο, το οποίο θα ήθελα να τονίσω, είναι το εξής. Ο γενικός μηχανισμός έδειξε ότι δεν, είναι, δεν λειτουργεί σωστά. Πολύ σπάνια έφτανε στην απόφαση μη επιστροφής. Αυτό είναι κάτι που ίσως θα μπορούσε να συζητηθεί αργότερα. Όσον αφορά την πρόταση αυτή καθε αυτή, καθορίζει προθεσμίες, το είπα αυτό ήδη και αυτό είναι πολύ καλό. Επίσης είναι καλό ότι έχει συγκεκριμένους ε, κανόνες δικονομικούς παρόλο που το είχαμε αυτό στην εσωτερική νομοθεσία καλύτερα να αναφέρονται άμεσα στον κανονισμό, διότι αντικατοπτρίζονται έτσι βέλτιστες πρακτικές που έχουν χρησιμοποιηθεί από τα κράτη-μέλη, ειδικού κανόνες και διατάξεις περί διαδικασιών επιστροφής που θα μπορούσαν να βοηθήσουν και να διευκολύνουν το έργο των δικαστών ίσως να παρέχουν μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου όσον αφορά τις διάφορες φάσεις της διαδικασίας επιστροφής και όσον αφορά τον ευρύτερο το γενικό μηχανισμό προβλέπονται κάποιες αλλαγές τα έγγραφα τώρα θα πρέπει να δίδονται με μετάφραση έχω κάποιες αμφιβολίες κατά πόσο αυτό αρκεί όσον αφορά το βασικό μηχανισμό κλείνοντας Ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι. Βασικά, το μεγαλύτερο, το πιο σημαντικό ζήτημα είναι κατά πόσο τα κράτη-μέλη και οι αρχές των κρατών μελών πραγματικά θα εφαρμόσουν πλήρως τους κανόνες συμπεριλαμβανομένων των προθεσμιών. Αυτό είναι το μεγαλύτερο ερωτηματικό που θέτω. Πώς θα δώσουμε κίνητρα στα κράτη-μέλη, ούτως ώστε να σέβονται τα κράτη-μέλη τους κανόνες. Πώς θα τα παρακινήσουμε. Κάποια από τα μέτρα θα πρέπει να διευκρινιστούν περαιτέρω. Ίσως βέβαια μιλούμε για κάποιες διακοσμητικές αλλαγές της διατύπωσης. Ίσως θα μπορούσαμε να εμβαθύνουμε και να ενισχύσουμε τους προτινόμενους μηχανισμούς και θα πρέπει να υπάρχουν και μηχανισμοί ασφαλείας όσον αφορά την άμεση συνεργασία κρατών μελών και φορέων των κρατών μελών τονίζεται κάτι καινούριο, ότι τα κράτη-μέλη μπορούν να συνεργάζονται με εξωτερικές κεντρικές αρχές. Αυτό μπορεί να είναι παρακινδυνευμένο όσον αφορά τη διαβίβαση πληροφοριών. Θα πρέπει να υπάρχει μια υποχρέωση κοινοποίησης, τουλάχιστον αυτό, κοινοποίησης προς τις κεντρικές αρχές, ούτως ώστε να είναι πλήρω ενήμερες οι κεντρικές αρχές για τα τεκτενόμενα. Άλλα άρθρα όπως το άρθρο 15, ίσως να πρέπει να διευκρινιστούν περαιτέρω, διότι πολύ συχνά τα δικαστήρια εφαρμόζουν τους κανόνες με διαφορετικό τρόπο. Και αυτό είναι κάτι που μπορεί να περιπλέξει μια υπόθεση και να την καθυστερήσει. Το σημαντικότερο, λοιπόν, είναι το εξής. Η νέα πρόταση παρουσιάζει κάποια ελπίδα, ελπίδα για βελτίωση όσον αφορά τη διαμεσολάβηση, ελπίδα όσον αφορά την αύξηση των συμμετοχικών δικαιωμάτων, αλλά ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι η de facto εκπλήρωση των υποχρεώσεων από πλευράς κρατών μελών. Και εξακολουθούν να υπάρχουν και κάποια περιθώρια αλλαγών και βελτιώσεων, όπως για το άρθρο 15. Βέβαια, θα καλωσορίσω οι εσδήποτε ερωτήσεις εκ μέρους σας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Φρίντρις και θα δώσω το λόγο τώρα στην Ανέτ Ολάντ, ανώτερη δικαστή στην Ολλανδία, θα μας πει ποια είναι η εμπειρία της όσον αφορά τη λειτουργία του μηχανισμού συνεργασίας. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Άκουσα τόσο πολλά θέματα, τόσο πολλές ενδιαφέρουσες απόψεις, έχω πάρα πολλά να πω, θα ήθελα μάλλον να πω πάρα πολλά για την διαμεσολάβηση, για τον μηχανισμούς, αλλά θα παραμείνω στον ρόλο μου ως δικαστού και θα αναφερθώ στις ε, δικαστικές ε, ανακοινώσεις και έχω υπόψη μου διαφορετικές χώρες. Ένα από τα τελευταία παραδείγματα είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά με το Brexit ε, δεν νομίζω να μας απασχολήσει ιδιαίτερα εντός του κανονισμού <clears throat> και θα προσπαθήσω να αποδείξω πως ε, η απευθείας επικοινωνία μπορεί να λειτουργήσει ως ε, να είναι αποτελεσματική. Έχω κάποιες ε, φωτογραφίες να σας δείξω, κάποιες στην οθόνη και θα σας πω πως ε, ε, μια οικογένεια που ένα Άγγλος Ολλανδί ζούσαν στην Αγγλία και μετά χωρίσανε. Όταν μιλάτε για απαγωγή τέκνου Συχνά όμως συμβαίνει ότι η μητέρα από την Ολλανδία κατοικεί στην Βασίλειο, δεν αισθάνεται καλά, θέλει να επιστρέψει στην χώρα της και προσπαθεί να δημιουργήσει μια νέα ζωή μετά από τον χωρισμό. Τα πράγματα δεν είναι πλέον όπως ήταν όταν ζούσαν μαζί επιστρέφει στην ε, Ολλανδία και παίρνει τα παιδιά μαζί της αλλά ο σύζυγος ε, διαφωνούσε. Τι, τι μπορεί να συμβεί λοιπόν και τι συνέβη στην περίπτωση. Δεν ήταν η Βασίλειο, ήταν μια άλλη χώρα, αλλά δεν έχει σημασία. Αυτό που συνέβη είναι ότι μετά από δύο δικαστικές ε, υποθέσεις οι οποίες εκκρεμούσαν στην κατοχώρηση και στον Βασίλειο για την ίδια υπόθεση φυσικά. Δεν λειτουργεί τώρα το μηχανάκι μου. Θέλω να μετακινηθούμε στην άλλη διαφάνεια. Τώρα, ο κανονισμός Βρυξέλλες 2, α, οι διαδικασίες ε, που αφορούν μια οικογένεια η οποία μπορεί να ε, κρεμοδικεί σε δύο χώρες και τα δύο, δικαστήρια μπορούν να λάβουν απόφαση αλλά μπορεί να μην συμπίπτουν οι απόφασεις και είναι εκτελεστή και στην άλλη χώρα αυτή η απόφαση. Το αποτέλεσμα λοιπόν ποιο είναι. Τι συμβαίνει εδώ πέρα. Σε αυτό το παράδειγμα ο δικαστής ε, στις κάτω που ασχολείται με το ζήτημα της απαγωγής δηλαδή κατά πόσον τα τέκνα θα πρέπει ή όχι να επιστρέψουν στο Βασίλειο. Και αυτός ο δικαστής ε, ε, διατάσσει την επιστροφή και τα τέκνα μετακινούνται στο Ινωμένο Βασίλειο. Αν ε, είναι άμεσα εκτελεστή, αυτό σημαίνει ότι τα παιδιά αρπάζονται θα λέγαμε από την αστυνομία, από τη μητέρα και μεταφέρονται στο Ινωμένο Βασίλειο. Στην πράξη όμως τα πράγματα μπορεί να είναι ακόμα χειρότερα. Ήδη τώρα έτσι που τα διηγούμε δεν είναι διόλου ευχάριστα. Μετά όμως ταυτόχρονα λίγο αργότερα, λίγο νωρίτερα ο δικαστής του Ενού λαμβάνει και αυτός μια απόφαση και ενδεχόμενα ο δικαστής αποφασίζει ότι τα παιδιά θα πρέπει να ζουν με τη μητέρα τους στις κατοχώρες αλλά ενταξύ τα τέκνα μπορεί να έχουν μετακινηθεί προς το Ηνωμένο Βασίλειο και αυτή βλέπουμε την κατάσταση εδώ στην φωτογραφία, στην ε, οθόνη. Βλέπουμε τους ε, Άγγλους ε, αστυνομικούς να παίρνουν τα παιδιά και να τα μεταφέρουν προς την Ολλανδία. Αυτό συμβαίνει όταν δεν υπάρχει επικοινωνία ανάμεσα στους δικαστές ή τις αρχές στα δύο κράτη-μέλη και έτσι οδηγούμεθα σε απόλυτη σύγχυση. Όχι, τόσο, όχι μόνο εμεί, αλλά και τα παιδιά και οι γονεί και οι υπολοιπε αρχέ. αρχές. Γίνεται ένα πινκ-πονγκ λοιπόν ανάμεσα στα κράτη-μέλη και αυτό είναι κακό για τα τέκνα αλλά και για του γονεί. Ε, όπως είπα σε αυτήν την περίπτωση υπήρξε άμεση επικοινωνία μεταξύ του δικαστηρίου στο ΙΤΑΒΙΤΑ και στι καλοχώρε. και ήρθαν σε επαφή, είτε ήσαν σε επαφή οι δικαστές, αρχικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ο Ολλανδός ε, συζητούσε με τον ε, Άγγλο, δικαστή, και αυτό συμβαίνει σε πολλές περιπτώσεις ε, επικοινωνούμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και όταν ε, ένα δικαστή θέλει να μιλήσει με, τον, με έναν συναδελφό του στην χώρα, μια άλλη χώρα, ναι, τότε ε, υπάρχουν και τα τηλέφωνα και σηκώνουν το τηλέφωνο και συζητάνε. Το Ολλανδικό Δικαστήριο είπε ότι έχουμε ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και θα αποφασίσουμε για θέμα της επιστροφής ή μη επιστροφής σε έξι μήνες. ο Ολλανδός ε, δικαστής είπε ότι εντός 6 εβδομάδων θα αποφασίσει. Θα κάνουμε λοιπόν μια κρόαση. μετά από τη λήψη της απόφασης. Ή 8 εβδομάδες περίπου μετά την απόφασή σας για να αποφασίσουμε εμείς το ΙΤΒ. Έτσι το δικαστήριο στο Μεγάλη Βρετανία είπε ότι η διαδικασία στην Ολλανδία διαρκεί 6 εβδομάδες. Άρα και σε εμά θα πρέπει να διαρκέσει 6 εβδομάδες. Και έτσι ο Ολλανδός ε, δικαστής ζήτησε να επιστραφούν τα παιδιά στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά είναι καλύτερο να περιμένουμε την εκτέλεση της απόφασης αφού το δικαστήριο στο Ηνωμένο Βασίλειο έλαβε την ε, απόφασή του. και μπορεί να καταστεί εκτελεστή μετά από έξι συν 2 εβδομάδες. Δεν υπήρξε επιβολή λοιπόν της απόφασης ε, μέχρι ότου να λάβει την απόφαση το δικαστήριο στο Ηνωμένο Βασίλειο και ε, ο Ολλανδός δικαστής είπε ότι και εμείς περιμένουμε την απόφαση του Αγγλικού Δικαστηρίου. Τα παιδιά λοιπόν μπορούν να περιμένουν στην Ολλανδία μέχρι να εκδοθεί η απόφαση στο Ηνωμένο Βασίλειο και να μην γίνεται αυτό το πινκ-πονγκ μεταξύ Ολλανδίας και Βασιλείου. Το θέμα είναι κατά πόσον θα πρέπει οι Ευρωπαίοι δικαστές να έχουν επαφή μεταξύ τους σε περιπτώσεις ε, απαγωγής σε άλλες ε, περιπτώσεις ε, διασυνοριακών υποθέσεων. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι το εξή. Πέρα από τη δουλειά μας, δηλαδή να ασχοληθούμε με τις ε, υποθέσεις, τα δικαστήρια, τις ακροάσεις και να λάβουμε αποφάσεις που χρειάζονται πολλές ε, διαδικασίες, χρειάζεται χρόνο, αλλά θα πρέπει να ε, ε, μπορούμε να ερχόμαστε και σε επαφή μεταξύ μας οι δικαστές. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα δίκτυο δικαστικό στην χώρα μας και το Ολλανδικό δίκτυο μας βοηθάει το να βρούμε ποιο είναι το αρμόδιο δικαστήριο ή ο αρμόδιος δικαστής το άλλο κράτος. Να ε. έρθουμε σε επαφή μαζί της ή μαζί του, με τι γλώσσα θα επικοινωνούμε και θα πρέπει να γνωρίσουμε ε, την ε, την γλώσσα, όπως καταλαβαίνετε, του άλλου κράτους. Όλοι έχουμε ένα δίκτυο υπό την αιγίδα της συνθήκης της Χάγης Θα πρέπει να έχουμε λοιπόν δικαστές εξειδικευμένους για θέματα ε, ε, οικογενειακού δικαίου. Αλλά θα πρέπει να υπάρχει και απαραίτητος χρόνος για να τη χάνουν και της σχετικής ε, στήριξης και αρρωγής. Λοιπόν, σας διαβεβαιώνω ότι σε κάποια κράτη-μέλη υπάρχουν δικαστές που χρησιμοποιούν το ιδιωτικό του email και κατηγορούνται από κάποιους ε, επειδή χρησιμοποιούν το ιδιωτικό του email και δεν, έχουν ασφαλή, δεν χρησιμοποιούν ασφαλές ηλεκτρονικό ταχυδρομείο από τα δικαστήρια και δεν τόσο ασφαλής η πληροφοριών και χρειάζεται γνώση και κατανόηση του κανονισμού οι δικαστές και εμπειρία του μηχανισμού στην πράξη. Ήδη το είπαμε, χρειάζεται εκπαίδευση, κατάρτιση επαγγελματικού τύπου συναντήσεις με άλλους δικαστές από άλλα κράτη-μέλη. Ε, προτείνα δύο κείμενα στην ε, ενημέρωσή μου που έκανα. Τώρα δεν είναι ενδιαφέρον να επαναλάβω αυτά που πρότεινα. Μπορείτε να διαβάσετε στο σημείωμά μου το ενημερωτικό. Αυτά και ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για αυτή την ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Έχουμε μερικά λεπτά για ερωτήσεις. Ε, ε, Ευχαριστώ πολύ. Ε, δεν έχω πολλές ερωτήσεις αυτή τη στιγμή, αλλά όλα αυτά τα πρακτικά προβλήματα τα οποία περιγράψατε δείχνουν πόσο σύνθετο είναι το θέμα αυτό και πόσο απολύτως αναγκαίο είναι για μας τους νομοθέτες να προβλέψουμε κάποιους μηχανισμούς που θα μας επιτρέψουν να γνωρίζουμε ποιο είναι το δικαιοδοτικό όργανο το οποίο είναι αρμόδιο για την εκδίκαση της υπόθεσης. Γιατί ε, είναι δυνατόν να ξεκινήσουν ε, διάφορες νομικές διαδικασίες σε διάφορες ε, χώρες, αλλά δεν είναι δυνατόν αυτό να αποτελέσει την καλύτερη δυνατή πρακτική. Θα πρέπει να γνωρίσουμε εκ των προτέρων ποια δικαιοδοσία θα ισχύσει και ποιο δικαστήριο θα επιληφθεί τη συγκεκριμένη υπόθεση. Και αυτό είναι εφικτό εφόσον υπάρχει αμοιβαία εμπιστοσύνη και αυτό προϋποθέτει ε, την ε, απαραίτητη νομοθεσία εκ μέρους των χωρών μελών και βεβαίως ε, προϋποθέτει και μια σωστή συνεργασία μεταξύ των κεντρικών αρχών ούτως ώστε να υπάρχει μια αμοιβαία ενημέρωση για όλα τα ενεχόμενα μέρη και μεταξύ των κεντρικών αρχών τόσο κατά την ε, προπαρασκευαστική διαδικασία αλλά και ε, κατά την τελική φάση της διαδικασίας όταν ε, η δικαστική απόφαση, η τιμιγορία θα πρέπει να εφαρμοστεί. Γιατί συχνά θεωρούμε ότι δεν υπάρχουν αρμόδια όργανα τα οποία να είναι αρμόδια για την εφαρμογή της δικαστικής απόφασης. Δεν είναι δυνατόν ένα παιδί να ε, το πάρει ένας ε, ε, υπάλληλο του δικαστηρίου για παράδειγμα και να το οδηγήσει στο... εκεί που έχει αποφασιστεί ότι θα πάει. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε μια ιδεώδη κατάσταση ε, που βεβαίως θα ήταν η εγγύηση των ε, καλών ε, συνθήκων για τη μελλοντική ανάπτυξη του παιδιού. Το όφελος του παιδιού δεν συμπίπτει πάντοτε με το συμφέρον των γονέων ή μια συγκεκριμένη χώρας το συμφέρον του παιδιού συνεπάγεται και την διατύπωση συγκεκριμένων κριτηρίων που ακριβώς θα εξασφαλίζουν τις ε, σωστές προϋποθέσεις. Εύελιν, ευχαριστώ πολύ. Εμένα με απασχολεί μία ερώτηση η οποία ε, ε, λανθάνει σε όλες τις συζητήσεις ε, τα λεγόμενα ε, ειδικά δικαστήρια τα οποία θα έπρεπε να συσταθούν. Και εδώ έχω ένα ερωτηματικό. Δηλαδή, ε, θα πρέπει να γίνει μια συγκέντρωση των αρμόδιων δικαστηρίων. Αυτό θεωρώ ότι είναι απολύτω εντάξει, όπω γίνεται στη Γερμανία, τη Γαλλία ή το Βέλγιο. Και αυτό είναι σωστό, γιατί ένας δικαστής ο οποίος μόνο μία φορά είχε μία τέτοια σχετική εμπειρία, δεν, έχει, δεν είναι δυνατόν να επιληφθεί αυτή τη υπόθεση. Η συγκέντρωση ναι, αλλά πρέπει να είναι ειδικά δικαστήρια ή είναι παρκές, φτάνει μάλλον τα υπάρχοντα οικογενειακά δικαστήρια να επιληφθούν αυτών των υποθέσεων, δηλαδή να μην συσταθεί μια ειδική δικαιοδοσία, αλλά τα ε, ήδη υπάρχοντα δικαστήρια να μπορούν να επιλαμβάνονται αυτών των υποθέσεων. Αυτό είναι το ζήτημα που με απασχολεί, γιατί δεν είμαι σίγουρη ε, για το τι ακριβώς ε, μιλάμε εδώ. Δύο πολύ σύντομες ερωτήσεις, λέει ο Πρόεδρος. Η πρώτη για τον κύριο Φρίντριχ. Οι αρχές της Τσεχίας, πόσες τέτοιες διασυνοριακές υποθέσεις αντιμετωπίζουν. Και ε, το παράδειγμα το οποίο μας έδωσε η κυρία Ολάντ ήταν παράδειγμα μιας βέλτιστης πρακτικής ε, συμβαίνει δηλαδή να μην υπάρχει επαφή μεταξύ των δικαστηρίων, δηλαδή ένα δικαστήριο να μην ε, γνωρίζει καθόλου ότι τη υπόθεση αυτή έχει επιληφθεί και ένα άλλο δικαστήριο σε κάποια άλλη χώρα. <laughs> Ο κύριος Φρίντριχ. Όσον αφορά τις ε, διασυνοριακές υποθέσεις, θα πρέπει να ορίσουμε πιο ξεκάθαρα τι είναι μια τέτοια είδους διασυνοριακή υπόθεση. Όσον αφορά τις απαγωγές απαγωνής, έχουμε 60-70 τέτοιες υποθέσεις το χρόνο απαγωγές στην Τσεχία 20-25 και οι υπόλοιπε είναι απαγωγές από την Τσεχία στο εξωτερικό. Και εδώ θα πρέπει να προσθέσουμε επίσης ε, υποθέσεις ε, ενώπιον των τσεχικών δικαστηρίων ε, τα οποία έχουν διασυνοριακά στοιχεία και τέτοιου είδου υποθέσεις μπορεί να φτάνουν μέχρι και τις 100 το χρόνο. Η κυρία Ολάντ. Η τελευταία ερώτηση ήταν μπορεί να συμβεί να μην υπάρχει καμία επαφή ε, μεταξύ δικαστηρίων και να εκκρεμούν ε, υποθέσεις σε δύο χώρες, η ίδια υπόθεση να εκκρεμεί σε δύο χώρες. Ναι, μπορεί να συμβεί, μπορεί να μην γνωρίζει το δικαστήριο ότι η υπόθεση εκκρεμεί σε μια άλλη χώρα. Και εάν δεν ε, αναφερθεί από τους γονείς, δεν δηλωθεί από τους γονείς, δεν μπορεί να το γνωρίζει το δικαστήριο ενδεχομένω. Είναι ευαίσθητο θέμα. Αλλά εάν ε, γνωρίζουμε ότι υπάρχει μία παράλληλη υπόθεση η οποία να εκκρεμεί σε μία άλλη χώρα, προσπαθούμε πάντοτε να έρθουμε σε επαφή και σας περιέγραψα τι γίνεται, είτε ετούμε την, ετούμεθα την μεταφορά της δικαιοδοσίας, ούτως ώστε να συνδυαστούν οι δύο υποθέσεις και να επαχθούν σε μία δικαιοδοσία, ε, προκειμένου να αξιολογήσουμε ποιο δικαστήριο έχει επιφυληθεί πρώτο της υπόθεσης. Εάν γνωρίζουμε ότι η υπόθεση κρεμεί σε μία άλλη χώρα, βεβαίως θα έρθουμε σε επαφή. Αλλά όπως είπα μπορεί να συμβεί να υπάρχει άγνοια. Και δυστυχώς όπως αναφέρθηκε πριν, ε, μερικές φορές ακόμα και μεταξύ κεντρικών αρχών Ε, όταν υπάρχει, όταν ε, ε, οι δικαστές έχουν επαφή μεταξύ τους με ένα email επικοινωνούν άμεσα. Αλλά άλλες φορές η επαφή αυτή μπορεί να γίνει μετά από εβδομάδες. Όταν ένα, εργασ... ένα δικαστήριο συγγνώμη, είναι αρμόδιο για μια υπόθεση, τότε τα πράγματα είναι απλά αλλά ε, όταν ε, οι γονείς απευθυνθούν σε διαφορετικά δικαστήρια, ε, τότε μπορούν να υπάρξουν πολλά προβλήματα. Και συμβαίνει να έχουν επιληφθεί δύο δικαστήρια επί τη βάση στοιχείων που τους έχουν ε, προσκομιστεί και θεωρώντας ότι είναι αρμόδια για την δικαιοδοσία. Είναι σημαντικό στο πλαίσιο της αναδιατύπωσης ακριβώς να αναφερθούν, να τα ζητήματα της μεταφοράς της δικαιοδοσίας. Βεβαίως θα πρέπει να υπάρχουν ε, βέλτιστες πρακτικές. Η βέλτιστη πρακτική να είναι αρμόδιο ένα δικαιοδοτικό όργανο, αλλά αυτό δεν ε, ανταποκρίνεται πάντως στην πραγματικότητα. Τότε θα πρέπει να γίνει η μεταφορά της δικαιοδοσίας και θα πρέπει να υπάρχει ένας τρόπος να διευθυνθεί το θέμα. Σας ευχαριστούμε. Ταντέρος θα πάρεις αμέσως το λόγο, αλλά πριν από αυτό Θέλεις να δώσεις κάποια απάντηση. Γιατί η κυρία Κρούγκερ κάτι θέλει να πει. Ταντέου, έχεις το λόγο. Θέλω να πω το εξής. Όσον αφορά την επιλογή της δικαιοδοσίας θα πρέπει να το εξετάσουμε. Μάλλον το εξετάσαμε αυτό το ζήτημα όταν ε, ασχοληθήκαμε με τον κανονισμό Ριξέλες 1, αλλά το ζήτημα των δικαιώματος του παιδιού δεν είναι αντικείμενο εμπορίου, δεν μπορούμε να το κάνουμε μια τέτοια σύγκριση. Φυσικά μπορούν να εκκρεμούν δύο η ίδια υπόθεση σε δύο κράτη-μέλη, αλλά ο κανονισμός θα πρέπει να συνταχθεί με τέτοιο τρόπο προκειμένου να καθίσταται σαφές ποια, ε, ποιο δικαστήριο είναι αρμόδιο και θα πρέπει να επιληφθεί τις υποθέσεις. Ο δικαστής Ποστούλσκι θα δείξει φυσικά το ζήτημα της κατάρτισης και εκπαίδευσης των δικαστών. Θα ήθελα να καταστεί σαφές το ποιο δικαστήριο είναι αρμόδιο σε ποια υπόθεση. Φυσικά είναι θέμα καλής ή ε, κακής θέλησης. Υπάρχει μια περίπτωση υπόθεση να εκκρεμεί σε μια χώρα και ε, ο άλλο κράτος να μην γνωρίζει το θέμα. Εάν η μητέρα ζει σε μια χώρα και ο πατέρας ή κάποια άλλη. Αλλά πώς γίνεται να μην, μπορεί να, να μην υπάρχει επικοινωνία. Υπάρχει σίγουρα ε, κακή βούληση. Ή οφείλονται στο ότι οι υποθέσεις ε, ξεκίνησαν σε διαφορετικό χρονικό διάστημα. αλλά θα πρέπει να ε, αποφασιστεί ποια χώρα, ποια δικαστήριο συγγνώμη είναι αρμόδιο. Τώρα θα απαντηθεί συντομία αυτή η απάντηση, διότι έχουμε και ένα επόμενο πάνελ και δεν έχουμε καν 45 λεπτά στη θέση μας. Ποιος θα απαντήσει στην ερώτηση της Εύελη, α, η Κομισιόν. Ναι, Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα απαντήσω στα γερμανικά. Δυστυχώ η συνάδελφό μου έπρεπε να πάει σε κάποια άλλη συνάντηση. Λέγομαι Ανδρέα Σόλτ. Είμαι εμπειρογνώμων στην ε, Κομισιόν και προηγουμένω ήμουνα ε, διευθύντρια στην ε, Κεντρική Αρχή τη Γερμανία. Απάντηση. Η Επιτροπή θεωρεί επαρκή πολιτικές η αρμοδιότητα να συγκεντρωθεί σε έναν συγκεκριμένο αριθμό δικαστηρίων. Ε, σε ορισμένες χώρες υπάρχουν οικογενειακά δικαστήρια αλλά παρόλα αυτά συγκεντρώθηκαν σε ένα αστικό δικαστήριο. Άλλες χώρες έχουν 500 δικαστήρια και τα πράγματα δεν λειτουργούν τόσο καλά. Ε, θεωρώ ότι είναι σημαντικό ο κάθε δικαστής να, ε, να αναλαμβάνει περισσότερες υποθέσεις και ούτω, ούτως ώστε να έχει περισσότερη, μεγαλύτερη εμπειρία. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να πω ότι είναι το άρθρο 32 που αφορά ακριβώς τη συγκέντρωση και όχι την εξειδίκευση των δικαστηρίων. Όσον αφορά τις παράλληλε διαδικασίες, βεβαίω ε, υπάρχει ένας κανόνας όταν η ίδια υπόθεση εκκρεμεί σε διαφορετικά δικαστήρια. Αλλά το πρόβλημα στο οποίο αναφέρθηκε συνάδελφος είναι όταν υπάρχουν συναφή θέματα ε, ε, ε, για το ίδιο παιδί ένα δικαστήριο είναι αρμόδιο για την επιστροφή του παιδιού και άλλο, αρμόδιο να είναι αρμο... και άλλο δικαστήριο είναι αρμόδιο για τα ασφαλιστικά μέτρα και άλλο δικαστήριο να είναι αρμόδιο επί της ουσίας. Εκεί υπάρχουν παράλληλες διαδικασίες που αφορούν όμως την ίδια υπόθεση. <laughs> E- Κοιτάξτε, πάμε αμέσως ε, στο τρίτο πάνελ. Θα εστιαστεί αυτό στις σχέσεις με τρίτες χώρες χωρίς εισαγωγή στα διδόκτωρα Κέρστιν Μπάρστ από τη Σύμβαση της Χάγης για το ιδιωτικό ε, δίκαιο, πηχεσιακό δίκαιο. Λοιπόν, θα αναφερθώ στην πρόταση για την αδιατύπωση του κανονισμού 2α. Είσαστε πολύ γρήγοροι, λέει η Πρόεδρος. Αν κάνετε και 11 λεπτά, εντάξει, δεν τρέχει τίποτα. Α, ωραία, κέρδισε ένα λεπτό. Σε σχέση με την σύμβαση της ΧΑΙΣΕΝ και τις άλλες συμβάσεις σχετικές, οι δύο συμβάσεις αποτελούν τμήμα μιας ομάδας τεσσάρων συγχρόνων διεθνών συμβάσεων για το κοινωνικό δίκαιο τη Χάγη που θέλουν να προστατεύσουν τα παιδιά σε δυσυνοριακέ περιπτώσει. Πέρα από τη σύμβαση του 1980 και τη 1996, η, η σύμβαση για την υιοθεσία του 1993 και του 2007 για την διατροφή των παιδιών και το πρωτόκολλο τη διατροφή που ανήκει στις βασικές συμβάσει Έχουμε τέσσερι συμβάσει δηλαδή τελικά. Αυτέ έχουν στόχο συντονισμού. Θέλουν συνεκτική διεθνή ένωμη τάξη προστασία των παιδιών και αυτό σε διάφορες συνορικές περιστάσεις. Πεδίο τώρα του κανονισμού Βρυξέλλες 2α. 2α θα πάω πιο σιγά. Πιο σιγά. Το πεδίο λοιπόν του κανονισμού Βρυξέλλες 2α αναφέρεται στην Διεθνή Ενώμη Τάξη και το ομώνυμο Προεδρείο μας εξέτασε δύο θέματα εν την προετοιμασία της παρεμβάσεως σε αυτό το εργαστήριο. Αν ο κανονισμός Βρυξέλλες 2α τροποποιήθηκε σύμφωνα με τις προτάσεις της αναδιατύπωσης και θα είναι συνεπής με τη διεθνή Τάξη που ισχύει σε παγκόσμιο επίπεδο ή όχι και τα πόσο επιτυχάνεται συντονισμός μεταξύ παγκοσμίου ενόμου τάξεως και των άλλων μέσων που ανέφερα. Δεύτερη ερώτηση που θέλω να απαντήσω θετικά σε αυτή. Η πρόταση να επιβεβαιώνει συντονισμένη εφαρμογή των σχετικών νομικών εργαλείων διευκρινίζει τη σύνδεση μεταξύ του κανονισμού Βρυξέλλες 2α και των συμβάσεων της Χάγης και συμβάλλει του τρόπο σε ασφάλεια δικαίου. Διευκολύνει του αξιωματόχου των κυβερνήσεων, δικαστέ, νομικού και άλλου φορεί να κατανοήσουν τη σχέση μεταξύ διεθνών νομικών μέσων σε κάθε περίπτωση. Εν συντομία, αναφερθώ σε κάποια σημεία. Δηλαδή, κατά πόσο ο κανονισμό Βρυξέλλε 2α συνάδει με το διεθνέ παγκόσμιο καθεστώ κυρίως με τις συμβάσεις 1996-1980. Δεν μου το είπε ο χρόνος να αναφερθώ σε λεπτομέρειες. Παρακαλώ, διαβάστε το έγγραφο του μονίμου Προεδρίου που προετοιμάσαμε για το εργαστήριο αυτό. Για περισσότερες πληροφορίες. Ευθύ εξ αρχής, σημειώνω ότι κάποιες διατάξεις θα και αναδιατύπωσή του θα οδηγήσουν σε διαφορές ανάμεσα στις δύο συμβάσεις. Πάντως, η Μολονότι πάνω τι διαφορέ δεν θα έχουν ερωτικέ επιπτώσει στην διεθνή ένωμη τάξη. Επίσης, γνωρίζουμε ότι κάποιε διατάξει ε, τη νέα πρόταση ε, αντιμετωπίζουν κάποιε προκλήσει που τα κράτη-μέλη γνωρίζουν σε σχέση με την ε, πρακτική εφαρμογή του κανονισμου βρυξελλε Βρυξέλλες 2α. Και κάποιες αυτέ τι προκλήσει έχουν σχέση και συγκρίνονται με τις δύο συμβάσεις ε, αντιμετωπίζουν το ζήτημα των ε, θέμητων καθυστερήσεων σε σχέση με τη διαδικασία επιστροφής των ε, εσφαλμένους απομακρυνθέντων τέκνων. 18 εβδομάδες είναι το περιθώριο για την επιστροφή. Η σύμβαση του 1998 υποχρεώνει τα κράτη-μέλη να ε, προβούν ε, άμεσα στις ε, διαδικασίες αυτές, αλλά να αναφέρει κάποιο χρονικό όριο, ενώ στο οποίο θα πρέπει να γίνει αυτή η μετακίνηση. Η σύμβαση του 1980 προβλέπει την δυνατότητα εφαρμογής κάθε δυνατού μέσου για να επιταχύνει τις διαδικασίες αλλά η ταχεία διαδικασία παραμένει μια πρόκληση για, σύμφωνα με τη διαδικασία του 1980. Οι τροπολογίες ότι φορά το χρονικό διάστημα για περιπτώσεις ε, απαγωγής ε, αναφέρουν ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστεί το ζήτημα και επίσης εδώ θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι μας θυμίζει το γεγονός ότι η θεμερίδα αρχή της σύμβασης του 80 ότι η επιστροφή θα προστατεύσει την ε, τέκνο από την ε, επιπτώσεις απαγωγής παρά μόνο εάν αυτή η επιστροφή γίνει τάχιστα. Μια άλλη προτινόμενη τροπολογία είναι η υποχρέωση των κρατών μελών να επικεντρώσουν τις υποθέσεις αυτές σε ε, περιορισμένο αριθμό δικαστηρίων. Περισσότερα από 40 συμβαλόμενα κράτη δημιούργησαν ε, ένα υψηλό ποσοστό ε, συνεργασίας και οδήγησαν στην αμοιβαία κατανόηση μεταξύ των βουλευτών και οδήγησε σε καλύτερη συνέπεια της ε, πράξης των δικαστών. Μια άλλη τροπολογία αφορά τα επίγοντα μέτρα για την προστασία του τέκνου. Ε, η πρόταση μπορεί να τύχει αναγνώριση στα κράτη στο οποίο βρίσκεται εγκαταστημένο το τέκνο. Το είναι ευπρόσδεκτη αυτή η τροπολογία διότι αφορά την προστασία διασυνοριακώς του τέκνου ε, σύμφωνα με την ε, σύμβαση του 86. Τώρα, <clears throat> οι αρχές ε, κάθε συμβαλόμενου κράτους θα πρέπει να έχουν δικαιοδοσία προκειμένου να αναλάβουν κάθε μέτρο προστασίας για το τέκνο και αυτά τα μέτρα έχουν εξωεδαφική ε, ισχύει. Το άρθρο 11 διασφαλίζει ότι ένα μέτρο προστασίας για την ασφαλή επιστροφή του απεχθέντος τέκνου θα επιβληθεί στο κράτος το οποίο το, κράτος, το τέκνο θα επιστραφεί. Και επίσης θα τύχει εγγύησης μέχρι ότου τα, οι αρχές λάβουν τα απαραίτητα μέτρα. Τώρα, η αναδιατύπωση αναφέρει ρητά πως το δικαστήριο σε μια παρόμοια απόφαση θα είναι υποχρεωμένο να την καταστήσει εφαρμοστή, εφαρμοστέα. Αυτό που είναι γεγονός είναι ότι αν οι διαδικασίες είναι τάχιστες ε, δεν θα ε, υπάρξει κίνδυνος ε, για το παιδί. Τα συμβαρόμενα μέρη έχουν υποχρέωση να ε, να εφαρμόσουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις προκειμένου αυτή η επιστροφή να γίνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την προστασία του τέκνου. Η διαταγή επιστροφής η οποία δεν είναι ε, τέλεση δίκη δεν θα έπρεπε να υπάρχει προκειμένου να μπορούμε να ανταποκριθούμε σε στις περιπτώσεις αυτές. Το Προεδρείο θεωρεί ότι αυτή η αναδιατύπωση αντανακλά αυτές τις ε, διατάξεις ε, χωρίς να επιβάλλει την υποχρέωση για, ε, σχετικά με την εκτελεστότητα της υπόθεσης, της απόφασης. Τέλος να επανέλθω στην διάταξη που λέει ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να φροντίσουν ότι οι κεντρικές αρχές έχουν τους επαρκείς πόρους για να προχωρήσουν στην εφαρμογή της απόφασης. Κεντρικές αρχές λοιπόν που έχουν οριστεί από τα συμπαλόμενα μέρη σήμερα με την οδηγία του 88 και του 96 διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο για την υλοποίηση της σύμβασης σε ειδικές συναντήσεις οι επιτροπές θα πρέπει να ενθαρρύνουν τις ε, κεντρικές αρχές και να τους προσφέρουν ε, το απαραίτητο οικονομικά μέσα αλλά και το απαραίτητο προσωπικό. Συχνά όμως αυτές οι αρχές δεν έχουν απαραίτητο προσωπικό και ε, χρήματα και έτσι η πρόκληση παραμένει. Το μόνιμο Προεδρείο ε, την ικανοποίησή του για αυτήν την αναδιατύπωση. Επίση, οι κεντρικέ αρχέ συνήθως ε, ε, συμπίπτουν με αυτές τις, ε, των 286 86 και 90. Διασφαλίζουμε ότι οι απαιτήσει αυτές θα πρέπει να έχουν θετικές συνέπειες προς όφελος της εφαρμογής αυτών των δύο συνθήκων, συμβάσεων. Να ολοκληρώσω λέγοντα ότι και άλλες τροπολογίες πιστεύουμε ότι έχουν θετικές επιπτώσεις. Τώρα το χρονικό διάστημα για την διευθέτηση υποθέσεων απαγωγής ή για την τοποθέτηση του και οι διατάξεις που προβλέπουν στην ενίσχυση και ενδυνάμωση της συνεργασίας ανάμεσα στις αρχές και τα δικαστήρια <clears throat> θα επηρεάσουν με θετικό τρόπο την εφαρμογή των οδηγιών του 1980 και του 1996. Λοιπόν, το μόνιμο Προεδρείο λοιπόν ε, καλωσορίζει τις αλλαγές στην, στην κανονισμό Βρυξέλλες 2α πάνω σε θέματα προστασίας των τέκνων. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστούμε πολύ και θα καλέσω άμεσα τον καθηγητή του Πανεπιστήμιου της Βαρκελών. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Για μένα είναι ικανοποιητικό το ότι παρεμβαίνω σήμερα για τέτοιου είδου θέματα, λαμβάνοντα υπόψη ότι τίθενται σαν ένα ερώτημα. Τι ε, γίνεται με τις ε, ε, με, τα προβλήματα αυτών των οικογενειακών διαφορών. Και στην πραγματικότητα θα έλεγα ότι η πρόταση από την Ευρωπαϊκή Ομάδα Ιδιωτικού Δικαίου ε, της οποίας προείσταμε έχει υποβάλει κάποιες ε, προτάσεις για τα ζητήματα αυτά. Στις περιπτώσεις αυτές ε, ε, βρισκόμαστε ενώπιον θεμάτων τα οποία πραγματεύεται η πρόταση αυτή. Και υπάρχει ένα πρόβλημα με το άρθρο 81 ε, της ε, Ευρωπαϊκής Συνθήκης, το οποίο απαιτεί ομοφωνία. Και θα, ενδεχομένως θα προκύψουν ε, διάφορες ενστάσεις εκ μέρους των χωρών μελών που είναι ευαίσθητα ως προς το θέμα αυτό. Τώρα, καταρχήν όσον αφορά το πεδίο εφαρμογή του κανονισμού, είναι η πρώτη δυσκολία και δεύτερη δυσκολία είναι τα κριτήρια ορισμού της αρμόδιας δικαιοδοσίας. Το πρώτο ερώτημα το οποίο θέτω είναι κατά πόσο ε, τα θέματα αυτά της ε, γονεϊκής ε, ευθύνης θα, θα πρέπει να επιλέγονται από το ίδιο όργανο. Γιατί με τον τρόπο αυτό μπορεί να υπάρξει, συγκεκριμένη, να υπάρξει κάποια σύγχυση εν σχέση με τι τροποποιήσεις θα πρέπει να γίνουν και ποια μέτρα θα πρέπει να διατερηθούν επί 20 χρόνια ε, το καθεστώς αυτό επίλυσης των ε, γονεϊκών διαφορών έχει παραμείνει το ίδιο. Ε, μέχρι στιγμής ε, υπάρχουν ζητήματα δικαιοδοσίας κλπ. Το δεύτερο ερώτημα στο οποίο δίδεται αρκετή προσοχή είναι και πόσο θα πρέπει να διατηρηθούν εντός του κανονισμού το ειδικό καθεστώς το οποίο προβλέπεται από το άρθρο 63. Στην Ισπανία υπάρχουν πολλές δυσκολίες ε, με, τα, με τη λειτουργία των εκκλησιαστικών ε, δικαστηρίων σε σχέση με τα αστικά δικαστήρια. Ε, και αυτό έχει κάποιες επιπτώσεις γιατί στο άρθρο 1 του κανονισμού αναφέρεται ότι πρόκειται για αστικά θέματα. Άρα στην περίπτωση αυτή θα έπρεπε να περιοριστεί το πεδίο εφαρμογής. Τρίτο ερώτημα. Το... Ο κανονισμός αναφέρεται ε, σε περιπτώσεις διαζυγίων ή χωρισμών αλλά παραμένουν εκρεμείς κάποιες, ε, κάποια ερωτήματα. Για παράδειγμα, τι γίνεται με τα διαζύγια ε, ομοφιλόφιλων ζεύγων. Ε, <laughs> ζευγών. Είναι μια πολύ δύσκολο να επιληφθεί η ερώτηση. Παρ' όλα αυτά είναι ένα πρόβλημα υπαρκτό. Δεύτερον, τι συμβαίνει με τα ιδιωτικά διαζύγια. Υπάρχει πρόταση της Επιτροπής ότι ε, εδώ, ότι στις περιπτώσεις αυτές δεν είναι, ε, δεν είναι αρμόδια τα δικαστήρια, υπάρχουν πολλές ε, φορές συμβολογράφοι οι οποίοι κάνουν τέτοιου είδους ε, ιδιωτικές συμφωνίες. Επίσης ε, υπάρχουν άλλα θέματα. Για παράδειγμα, η αναγνώριση στη Γερμανία ενός ε, διαζυγίου το οποίο έγινε στην Συρία σύμφωνα με τον Ισλαμικό νόμο. Άρα λοιπόν ε, γύρονται πολλά θέματα. Γιατί το ζητούμενο εδώ είναι να διευκρινίσουμε τι συμβαίνει με τέτοιου είδους ε, θέματα. Το τρίτο ερώτημα ε, σχετίζεται με την κύρωση του γάμου. Και εδώ υπάρχουν κάποιοι υπάρχει μια διαφορά μεταξύ ε, θα πρέπει να γίνουν κάποιες διακρίσεις. Εδώ ε, βλέπουμε ότι υπάρχει ε, μια εξέλιξη και πρόκειται για μια Διαδικασία ακύρωση Muchas cosas que decir sobre este, Τι γίνεται στις περιπτώσεις όπου αποβιώνει ο ένας από τους ε, δύο συζύγους. Και τώρα θα έρθουμε στο δεύτερο τμήμα που αφορά την ε, αρμοδιότητα των αρχών. Αυτό το οποίο εδώ ε, θεωρώ ότι χωλαίνει είναι ότι δεν αναφέρεται το ζήτημα της αυτόνομης βούλησης. Εάν θα θέλαμε, ε, αν η, Επιτροπή, η πρόταση Επιτροπής παρέπεμπε στην ε, συνθήκη της Ρώμης, το άρθρο 3α, ε, στην περίπτωση αυτή θα έπρεπε να επιλεγεί το εφαρμοστέο δίκαιο και θα μπορούσαμε όλοι να συμφωνήσουμε. Ωστόσο, ο κανονισμός αυτός έγινε δεκτός μέσω της διαδικασία της ενισχυμένη συνεργασία. Άρα δεν μπορούμε να αναμένουμε μια τέτοια είδου τροποποίηση. Το ζήτημα είναι κατά πόσο είναι δυνατόν να γίνουν αυτές οι διευκρινήσει και να συμπεριληφθούν εδώ. Όσον αφορά τώρα τα κριτήρια και το σκοπό του προσδιορισμού της ε, αρμοδιότητας. Εδώ η Κομισιόν αναφέρει 7 ε, κριτήρια τα οποία όμως δεν έχουν καμία συνοχή μεταξύ τους. Άρα λοιπόν υπάρχουν ε, κάποιοι κίνδυνοι εδώ και ενδεχομένως αυτό θα οδηγήσει σε, μια, σε έναν ανταγωνισμό μεταξύ των δικαιοδοτικών οργάνων και δεν διευκρινίζεται παρκώς ποιο δικαστήριο είναι αρμόδιο. Και όλα αυτά ισχύουν μέχρι σήμερα. Τώρα, όσον αφορά όλα αυτά τα κριτήρια, θα ήθελα να πω ότι το ζητούμενο δεν είναι να υπάρχουν περισσότερες ε, δυνατότητες λήψης αποφάσεων, αλλά το ζητούμενο είναι να υπάρξει μια ομοφωνία. Ε, το κείμενο αυτό καθ' αυτό, στο σύνολό του, βεβαίως εισάγει ορισμένα κριτήρια. Αλλά αυτό το οποίο εμείς ε, καλούμεθα να αξιολογήσουμε είναι μια... κατά πώς θα έπρεπε να γίνει μια ιεράρχηση εδώ. Γιατί δεν είναι δυνατόν ε, κάθε φορά να πρέπει να επιλέγει το αρμόδιο δικαιοδοτικό όργανο. Εάν ε, κάνουμε πράγματι μια τέτοια ιεράρχηση, στην περίπτωση αυτή θα πρέπει θα έχει αυτό και κάποιες συνέπειες όσον αφορά τις εναλλακτικές δυνατότητες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Ορισμένα άρθρα οδηγούν ε, σε σημαντικές ε, διαφωνίες. Το άρθρο 6 και το άρθρο 7. Το άρθρο 6 αφορά την αποκλειστική αρμοδιότητα, αλλά με την έννοια αυτή, αποκλειστική αρμοδιότητα, έχουμε ε, εδώ δίδεται μια εντελώ διαφορετική σημασία από ό,τι στον ε, κανονισμό Βρυξέλλες 2. Ε, Πιστεύω ότι η, πρόταση, ε, ότι η Κομισιόν εδώ προτείνει να διαγραφεί αυτή η διάταξη, αλλά στο άρθρο 7 θα έπρεπε να διατηρήσουμε την σκέψη να ε, συσταθεί ένα φόρουμ. Ε, πρόκειται για μια θετική σκέψη, αλλά θα πρέπει βεβαίως να γίνει εδώ μια διαφοροποίηση μεταξύ της, ε, του πεδίου εφαρμογής των κανόνων των χωρών μελών εάν δεν είναι ξεκάθαρο το ζήτημα της αρμοδιότητας σε ένα άλλο επίπεδο. Οι Ευρωπαίοι πολίτες θα πρέπει να μπορούν να είναι βέβαιοι ότι οι λύσεις και οι αποφάσεις για τις συζυγικές τους ε, κρίσεις και για τον προσωπικό τους ε, βίο ε, μπορούν να βρουν μια ικανοποιητική λύση. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν περισσότερα προβλήματα παρά λύσεις και δεν ξέρει κανείς με τι θα πρέπει να ταυτιστεί. Θα πρέπει βεβαίως θα πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές οι οποίες όμως είναι προφανείς και επί των οποίων είναι δυνατόν να υπάρξει μια ομοφωνία. Εάν δεν μπορούμε να πετύχουμε αυτή την ε, ομοφωνία στα επιμέρους σημεία, θεωρώ ότι θα έπρεπε να αφήσουμε τα πράγματα όσα έχουν. Αυτή είναι η άποψή μου για την πρόταση Επιτροπή. Uh, Ευχαριστώ κυρία καθηγήτρια. Τελευταίος, ο δικαστής Ποστούλσκι. Γενικός Γραμματέας του Ευρωπαϊκού Δικτύου Κατάρτισης Δικαστών. Έχετε το λόγο για ένα δεκάλεπτο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, μας δώσετε το λόγο. Ξεκινώ ευχαριστώντας τους οργανωτές που συμπεριέλαβαν στην ημερήσια διάταξη του εργαστηρίου το θέμα των, της των δικαστών. Αυτό το θέμα της δικαστικής κατάρτισης θεωρείται σαν βασικό εργαλείο που εξασφαλίζει ότι τα δικαιώματα που δίνει το ευρωπαϊκό δίκαιο μπορούν να γίνουν πραγματικότητα. Υπάρχει αυτή η σχέση που έχουμε δίπλα στο ερωτηματικό. Δηλαδή υπάρχει σχέση μεταξύ των μέσων του ευρωπαϊκού δικαίου και της δικαστικής κατάρτισης. Αναφέρθηκε η κατάρτιση από πάρα πολλούς ομιλητές σήμερα το απόγευμα, οπότε τουλάχιστον σε αυτή την αίθουσα υπάρχει γνώση για την ανάγκη της κατάρτισης. Είτε μιλάμε για ένα νέο εργαλείο είτε όχι. Δυστυχώς εκτός της αιθούσης αυτής ε, δεν είναι ιδιώδης ο κόσμος. Και η αύξηση της ευαισθητοποίησης για την ανάγκη κατάρτισης είναι ακόμα τεράστιο πρόβλημα για όλους τους φορείς. Ε, ε, για την δικαστική αυτή πολιτική που ακολουθούμε αυτά είναι σημαντικά για να πετύχουμε το αποτέλεσμα, αυτό που ζητά. Δεν αρκεί να είναι απλώς καλά διατυπωμένος ο κανονισμός και βελτιωμένος για το οικογενειακό δίκαιο σε συνορικό επίπεδο. Αυτό που είναι κρίσιμο είναι να έχουμε πρακτική εφαρμογή αυτών των διατάξεων. Και εδώ είναι θεμελιώδης ο ρόλος των εισαγγελέων, των δικαστών και άλλων εκπροσώπων του νομικού ε, κλάδου να εφαρμόσουν σωστά τις διατάξεις. Οι δικαστές θα πρέπει να μπορούν σωστά επαγγελματικά δεόντως να εκτελούν τα καθήκοντά τους, συμπεριλαμβανομένων των καθηκόντων στα πλαίσια της ευρωπαϊκής νομοθεσίας πρέπει να έχουν επαγγελματικές δεξιότητες. Και όταν οι δικαστές εμείς διορίζουμε δεν ε, τελικά διαφωτιζόμεθα λόγω διορισμού. Θα πρέπει να αποκτήσουμε τις ε, επαγγελματικές δεξιότητες ε, και κυρίως μέσω κατάρτισης και αυτό ισχύει κυρίω όταν έχουμε νέα νομικά μέσα. Και αυτή η αναδιατύπωση Βρυξέλλες 2α είναι ένα τέτοιο εργαλείο, χρειάζεται ε, εκτεταμένες ε, εκπαιδευτικές δραστηριότητε. και όπως θα βλέπετε και στην οθόνη εντοπίζω τρεις βασικούς στόχους ε, τέτοιων διαδικασιών κατάρτισης. Πρέπει να γνωρίζουν οι δικαστές ότι υπάρχει με τη διαδικασία κατάρτισης. Δεν μπορούν να ξυπνήσουν χρόνια και μήνες μετά τη θέση σε ισχύ του μέσου όταν αντιμετωπίζουν μια υπόθεση και να δουν ότι έπρεπε να έχουν τη γνώση. Θα πρέπει να προετοιμαστούν, να το γνωρίζουν ότι μπορεί να υπάρξει κατάρτιση, πρέπει να προετοιμαστούν, αυτό είναι το δεύτερο σημείο, να αυξήσουν τι γνώσει του, τι δεξιότητές του, θα μπω σε λεπτομέρειες αργότερα, τι δεξιότητε απαιτούνται, τι είδου γνώση απαιτείται, ούτω ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν. Και τρίτον, οι δικαστέ θα πρέπει να είναι αφοσιωμένοι, να θέλουν να πετύχουν τους στόχους του μέσου. Θα πρέπει να πιστεύουν ότι που εκτελούν σημαντικότητα καθήκοντα εφαρμόζοντας ορθώς το εργαλείο που υιοθετείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητε και σωστή τομεί είναι προπετούμενα, είναι απαραίτητα. Οι δραστηριότητε κατάρτιση θα πρέπει να λάβουν χώρα σε δύο επίπεδα, σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό. Υπάρχει τεράστια διαφορά στο τι μπορεί να επιτευχθεί σε κάθε από τα δύο επίπεδα. Θα ήθελα, εν συντομία, να παραθέσω τους τομείς στους οποίους απαιτείται η κατάρτιση. Αλλά πριν από αυτό θέλω να παρουσιάσω ακροθυγώς τι προσφέρεται στο διασυνοριακό οικογενειακό δίκτυο. Θα το παρουσιάσω από πλευρά του Ευρωπαϊκού ε, Δικτύου ε, Καταρτήσεως Δικαστών. Το δίκτυο είναι αρκετά δραστηριοποιημένο στην παροχή κατάρτισης στον τομέα διασυνοριακού οικογενειακού δικαίου. Να σας υπενθυμίσω ότι το EGTN είναι δίκτυο 35 εθνικών φορέων κατάρτισης των 28 κρατών μελών στην Ακαδημία του Ευρωπαϊκού Δικαίου. Τι κάνουμε εκτελούμε δραστηριότητε σε ευρωπαϊκό επίπεδο και προσπαθούμε να ανταλλάξουμε και απόψει μεταξύ εθνικών φόρεων, τεχνογνωσία. προς να κινούμεθα καλύτερα και σε εθνικό επίπεδο. Τρίτο τρόπο, οργανώνουμε διάφορε μορφέ κατάρτιση με διαφορετικά θέματα. Βλέπετε τον κατάλογο με σεμινάρια, ανταλλαγές, ε, γλωσσική εκπαίδευση, δραστηριότητε που αφορούν τους ερχόμενου στο επάγγελμα, του μελλοντικού εισαγγελεί και δικαστέ αυτούς που περνάνε από την βασική εκπαίδευση. Στον τομέα διασυνοριακού οικογενειακού δικτύου ετησίως διοργανώζουμε σεμινάρια, σεμινάρια που εστιάζονται επί του κανονισμού Βρυξέλλες 2α, αλλά προσπαθούμε να εστιάσουμε και τα σεμινάρια μας και επί διαφόρων υποθέσεων. Μελετούμε μαζί με τους μετέχοντες σεμινάρια διάφορες υποθέσεις, πρακτικά παραδείγματα, βέλτιστες πρακτικές σε διασυνορική συνεργασία μεταξύ δικαστηρίων, μεταξύ δικαστηρίων και εθνικών αρχών. Πέρσι εστιαστήκαμε και στο πώς μπορούμε να προσεγγίσουμε τα παιδιά, πώς να ακούμε τα παιδιά, πώς να προστατεύουμε τα δικαιώματα των παιδιών. Αυτά τα σεμινάρια έχουν σαν στόχο την εμβάθυνση των γνώσεων των συμμετεχόντων σε τέτοια σεμινάρια περί ευρωπαϊκών μέσων. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί και σε εθνικό επίπεδο, σε τέτοια κατάρτιση. Ποια είναι η προστιθεμένη ε, αξία των σεμιναρίων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πάρα πολλά πλεονεκτήματα. Πρώτα απ' όλα, όταν οι δικαστές συναντώνται, μπορούν να ανταλλάσσουν εμπειρίε με του δικαστέ από άλλο κράτο μέλο Ευρωπαϊκή Ενώσεω, μπορούν να συναντήσουν Ευρωπαίου εμπειρογνώμων να συζητήσουν μαζί του. Μπορούν να το κάνουν και σε ξένε γλώσσε, οπότε βοηθά να μάθουν ξένε γλώσσε και δημιουργούν δίκτυα. Αυτά τα προσωπικά δίκτυα τα οποία αναφέρθηκαν εδώ, που είναι ακρογωνιαίο λίθο τη αμοιβέ εμπιστοσύνη μεταξύ του τα προγράμματα αυτά ανταλλαγών που έχουμε οργανώσει σε επίπεδο EGTN επί 10 χρόνια κατ' το λέει του Ευρωκοινοβουλίο Είναι ο καλύτερο τρόπο οικοδόμηση αμοιβέ εμπιστοσύνη. Στέλνουμε για δύο εβδομάδε δικαστέ σε ένα άλλο κράτο μέλο. Συνεργάζονται με ένα ομότιμό του, ε, ασχολούνται με υποθέσει από κοινού και βλέπουν πώ οι ίδιε οι καταστάσει προσεγγίζουν του δικαστέ σε ένα άλλο κράτο μέλο και σε άλλο εθνικό δίκαιο. Βέβαια, τους εκπαιδεύουμε και σε γλώσσες για να μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτές τι εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε ξένες γλώσσες να μπορούν να παρακολουθήσουν και να μάθουν το ευρωπαϊκό δίκαιο. Διοργανώνουμε τα προγράμματα για τους νοδιοριστέντες δικαστές. Δεν θέλω να παρουσιάσω τώρα και τον διαγωνισμό που περιγράφεται στο ενημερωτικό μου σημείωμα. Αυτά λοιπόν προσφέρονται ευρύτατη προσφορά ε, δραστηριοτήτων καταρτήσεως. Προσφέροντα αυτέ τι δραστηριότητε, βλέπουμε και πόσα προβλήματα και προκλήσει υπάρχουν. Προσπαθούμε να προσελκύσουμε του δικαστέ να συμμετάσχουν στι δραστηριότητε. Είδαμε μια πολύ καλή εικόνα τη Ολλανδή συναδέλφου με τον δικαστή που καθόταν ε, μπροστά σε ένα σωρό υποθέσεων. Ο φόρτο εργασία των δικαστών πράγματι είναι τεράστιο εμπόδιο. Δεν μπορούν να συμμετάσχουν εύκολα σε, σε κατάρτιση. Και αν βρουν χρόνο, έτσι επιτρέπουν οι ανώτεροι του να πάνε σε αυτά τα προγράμματα ανταλλαγή ή κατάρτιση. Αυτό είναι το πρόβλημα. Έχουν περιορισμένε γλωσσικέ γνώσει. Υπάρχει πρόβλημα έλλειψη εξειδίκευση των δικαστών. Αν πρέπει να επιλέξουν, αν θα πάω να κάνω κατάρτιση εθνικό δίκαιο, ευρωπαϊκό δίκαιο, που να ακούσω μία υπόθεση μία φορά το χρόνο, δύο φορέ το χρόνο, ποτέ δεν θα επιλέξουν την κατάρτιση όσον αφορά το ευρωπαϊκό δίκαιο και τα μέτρα λιτότητας σε κράτη-μέλη. Πολλά μέλη του EGTN περιορίζουν τους πόρους τους, οικονομικούς πόρους, ανθρώπινους πόρους. Ακόμα και αν υπάρχει προσφορά κατάρτισης δεν μπορεί να απορροφηθεί η προσφορά. Δεν υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι μπορούν να φιλοξενήσουν τις δραστηριότητες επίσης κατάρτισης. Υπάρχουν πολλά προβλήματα όσον αφορά τη διοργάνωση δραστηριοτήτων κατάρτισης. Τι να κάνουμε λοιπόν, πώς να το προσεγγίσουμε για να μπορέσουμε να προετοιμάσουμε τους δικαστές, τους εθνικούς δικαστές, ώστε να εφαρμόζουν τον αναδιατυπωμένο κανονισμό για το οικογενειακό δίκαιο. Πρώτα απ' όλα, όπως ε, είπα, πρέπει να γίνουν βήματα σε δύο επίπεδα. Ευρωπαϊκό, όπως το EGTN, όπως η Ακαδημία Ευρωπαϊκού Δικαίου από το TRIER, θα πρέπει να οργανώσουμε περισσότερες δραστηριότητε αλλά θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τα εθνικά μέλη, τα μέλη μας στους εθνικούς φορεί εκπαίδευση να στέλνουν δικαστέ δραστηριότητε και να διοργανώνονται και δραστηριότητε σε εθνικό επίπεδο. Πρέπει να θυμόμαστε ότι πλευρά εθνική πάντα υπάρχει και μια ανάγκη επιλογή. Θα οργανώσω μια κατάρτιση για το δικό μου εθνικό δίκαιο ή θα αφιερώσω χρόνο και πόρου για κατάρτιση σε ευρωπαϊκό δίκαιο. Κάτι που δεν το βλέπω ότι είναι τόσο μεγάλη ανάγκη από την πλευρά της καθημερινής μου δουλειάς. Και από τις δύο πλευρές βλέπουμε ότι υπάρχει μια ανάγκη δραστηριοτήτων για να υπάρξει επιστητοποίηση, δηλαδή να, ότι υπάρχει ένα νέο εργαλείο και τι περιέχει αυτό το νέο εργαλείο. Πρέπει να υπάρχει γνώση γι' αυτό. Υπάρχει μια ανάγκη επίσης για αύξηση εμπιστοσύνης μεταξύ δικαστών, μεταξύ εθνικών συστημάτων, μέσω της διοργανώσεως περισσότερων ανταλλαγών. Αυτό μας οδηγεί βέβαια σε συγκεκριμένες εκπαιδευτικές ανάγκες που βλέπετε στην οθόνη, ανάγκες κατάρτισης. Και φτάνω τώρα στο τέλος του χρόνου μου, ένα λεπτάκι θέλω, άπειτα. Είμαι απελπισμένη, λέει ο Πρόεδρος, διότι μας τελειώνει ο χρόνος. Ο Ταντέους ξέρουμε ότι θα συναγάγει τα συμπεράσματα, μετά έχουμε ερωτήσεις και απαντήσεις, πρέπει να επιταχύνεται. Να επιταχύνεται λοιπόν, μισό λεπτό. Λοιπόν, βλέπετε λοιπόν, ότι αυτό το μισό λεπτό έχω στη διάθεσή μου, οπότε τι πρέπει να κάνω, πρέπει να συνοψίσω. Σα καλώ διαβάστε λοιπόν ε, το ενημερωτικό μου σημείωμα και θα δείτε στο ενημερωτικό σημείωμα ποια είναι τα σημεία τα οποία θέλουμε να εξετάσουμε και ποια πρέπει να επεξεργαστούμε, τόσο ώστε να κινηθούμε σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και να υπάρχει σωστή κατάρτιση των δικαστών και να εστιαστούμε από αυτού. Και επειδή δεν ε, ανησυχώ αν φορεί όπω το EGTN ή άλλοι φορεί ευρωπαϊκοί που παρέχουν κατάρτιση ότι θα τα στερνιστούν, Δεν ανησυχώ, θα δανώσουν κατάρτιση. Αλλά βλέπω τεράστια προβλήματα στο βαθμό στον οποίο θα γίνει αυτό σε εθνικό επίπεδο σε αυτό το τομέα. Αυτό με προβληματίζει. Όλε οι προσπάθειε από πλευρά των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων θα πρέπει να γίνουν σε αυτό το επίπεδο. Οι εμπλεκόμενοι στον εθνικό τομέα, στο εθνικό επίπεδο, οι εμπλεκόμενοι φορεί να γνωρίσουν ποιε ανάγκε υπάρχουν. Αυτές περιγράφονται οι ανάγκες πάρα πολύ ε, αναλυτικά στο ενημερωτικό σημείωμα. Είμαι ένα πάρα πολύ γενναιόδορη, λέει η πρόεδρος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεισφορά σας. Ελπίζω κανείς να μην έχει ερώτηση, λέει η πρόεδρος. Εκτός αν είναι κατεπήγον, Εύελιν, όχι, θα δέω. Έχεις το λόγο λοιπόν για να συναγράψει συμπεράσματα, θα δε. Λοιπόν, σε ευχαριστώ. Άκουσα, άκουσα όλο το σεμινάριο και για μένα πρέπει να πω ότι ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα αυτά που άκουσα και ευχαριστώ όλους τους ομιλητές μας. Θα μπορούσαμε, ίσως θα έπρεπε να έχουμε περισσότερο χρόνο για κάποια θέματα, αλλά ένα απόγευμα είναι σύντομο, τι να κάνουμε. Ε, και ήταν και πληρέστατο, πληρέστατο. Αλλά ήταν και έξοχο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, θα δε. Αυτό είναι το συμπεράσμά μου. Αλλά τώρα μπες εσύ στο ψητό. Ε, ευχαριστώ πολύ. Τα συμπεράσματά μου είναι τα ίδια. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους φιλοξενούμενους μας, όλους τους επαείοντες για τη δυνατότητα να εξετάσουμε τον όλο τομέα από διάφορες οπτικές γωνίες. Αυτό είναι κάτι που εμπλουτίζει τις γνώσεις μας. Πριν μπούμε στη σκληρή νομοθετική διαδικασία που πρέπει να ξεκινήσουμε και να πραγματοποιήσουμε στο Ευρωκοινοβούλιο. Επίσης, γινόμαστε πιο ευαίσθητοι ε, όσον αφορά τις κρίσιμες στιγμές που αφορούν την αναδιοτύπωση του κανονισμού. Τα περισσότερο ευαίσθητα ζητήματα σχετίζονται με την ειδική αντιμετώπιση της οποίας πρέπει να τύχει ένα παιδί. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ουσιαστικά έχει αφήσει εκτός όλες τις υποθέσεις οικογενειακές και τα προβλήματα του γάμου, αν θέλετε, συγκεντρωνόμαστε μόνο επί των γονικών ευθυνών και επί των διασυνοριακών απαγωγών. Μέχρι τη σημερινή, μετά τη σημερινή ακρόση, μάλλον συγγνώμη, είμαστε σίγουροι για ένα πράγμα, ότι δεν θα πρέπει να κάνουμε τίποτα το οποίο θα, θα επιδεινώσει την κατάσταση Um, όσον αφορά τον κανονισμό Βρυξέλλες 2 α. Το ίδιο ίσχε και με τις Βρυξέλλες 1. Βέβαια το αντικείμενο του κανονισμού ήταν διαφορετικό, όμως ε, πολλοί νομικοί μηχανισμοί μοιάζουν και κατά πολύ. Αυτό θα είναι το σύνθημά μας. Δεν θέλουμε να επιδεινώσουμε την κατάσταση, θα είναι το σύνθημά μας. Συμφωνώ και με την καθηγήτρια που πήρε το λόγο από την Ισπανία, δεν μπορούμε, αν δεν συμφωνήσουν όλα τα κράτη-μέλη, είναι καλύτερα να μην κάνουμε τίποτα. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ Βρυξελών 2 και Ρώμης 3. Στη Ρώμη 3 μπορούσαμε εύκολα να αποφασίσουμε επί των διαδικασιών της διευρυμένης συνεργασίας και δεν συνέβαινε κάτι φοβερό. Επτά κράτη-μέλη συμμετείχαν, άλλα κράτη-μέλη αποφάσισαν να μην συμμετάσχουν. Όμως η δυνατότητα επιλογής δικαιοδοσίας είναι δυνητική. Δεν είναι κάποια υποχρέωση. Όποτε ένα ζευγάρι παντρεύεται, έχει το δικαίωμα σε περίπτωση διαζυγίου. Το ζευγάρι λοιπόν έχει τη δυνατότητα να επιλέξει μια συγκεκριμένη δικαιοδοσία. Όμως δεν είναι ελεύθερη επιλογή, βασίζεται αυτή η επιλογή επί κάποιων ε, προδιαγραφών, ε, επί κάποιων περιοριστικών στοιχείων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Στην περίπτωση των Βρυξελών 2α θα πρέπει να συζητήσουμε επίσης παρόμοια στοιχεία. Για μία ακόμη φορά λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ για όλα σας τα σχόλια, ευχαριστώ για τη συζήτηση διότι αυτό με βοηθά πολύ ως εισηγητή, αλλά και τους συναδέλφους μου από την Επιτροπή. Γνωρίζω ότι θα παλέψουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα έχουμε πιθανότατα διαφορετικές απόψεις σε σχέση με το Συμβούλιο, αν συγκρίσουμε το Συμβούλιο, όμως αν θέλουμε να καταλήξουμε σε ένα αίσιο φινάλε, αίσιον πέρας, σίγουρα θα τα καταφέρουμε και είμαι βαθιά πεπισμένος